Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την συνήθη ανακοίνωση ότι λόγω και του απορρίτου σας ε, λέγω ότι θα υπάρχει κινηματογράφηση και μαγνητοσκόπηση της ε, ε, Συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα έγκριση τη μερισσία διατάξεως. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει, επομένως εγκρίνεται. Σημείο 2 αφορά τις ανακοινώσει του Προέδρου. Έχω να σα πω τα εξή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ένταξης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση για την ε, Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Πρέπει να σας πω ότι στην επόμενη Δευτέρα 17, ή μάλλον όχι, την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου ε, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, θα ξεκινήσουν ε, μαζί με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, στις 15 και 30 μέχρι τις 16 και 30. Εμείς θα ξεκινήσουμε την κανονική μας συνεδρίαση σαν αύκο την ίδια μέρα, αλλά θα ξεκινήσουμε στις 16 και 30. Ακριβώς έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την κοινή συνάντηση με τους διαπραγματευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όσον αφορά την συνεδρίαση ΚΟΖΑΚ, η υποκυπριακή προεδρία ε, υπήρξε μια συνάντηση της ε, ΚΟΖΑΚ και στις 17 Δεκεμβρίου 16 και 45 θα ξεκινήσει ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά το θέμα αυτό. Επίσης στις ανακοινώσεις έχω να σας πω ε, την παρούσα κατάσταση όσον αφορά τις διαδικασίες επικύρωσης ε, όπως ήθιστε κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και για την οικονομική διακυβέρνηση και για την ένταξη της Κροατίας. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, επομένως με 3 έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 5 Σεπτεμβρίου 2012. Είναι στη διάθεσή τα πρακτικά αυτά. Εάν δεν έχετε σχόλια ή αντιρρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα και τα πρακτικά και μπορούμε να περάσουμε επομένως στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως, το οποίο αφορά ή μάλλον να πω στα επόμενα δύο σημεία της ημερησίας διατάξεως είναι το καθεστώς και χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ιδρυμάτων. Η κυρία Γιαννάκου είναι η συγγήτρια. Ε, και επίσης την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, θέμα για το οποίο η είναι ο συνάδελφό μα Γκερέρο. Θα συζητήσουμε λοιπόν από κοινού τα δύο αυτά θέματα, αλλά βεβαίως πρώτα θα ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει σήμερα η, εισηγήτρια κυρία Γιαννάκου. Δυστυχώ, τα έγγραφα είναι στη διάθεσή σα μονάχα στα αγγλικά. Ξέρετε ότι η Επιτροπή Γιούρη είχε ζητήσει την εφαρμογή του άρθρου 50, αλλά τελικά άλλαξε γνώμη γιατί επιτύχαμε συμφωνία στην κοινή συνάντηση, επομένως απεσύρθη το αίτημα αυτό, όμως εν τέλει συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να αναβάλουμε την έγκριση της ε, ε, έκθεσης Γιαννάκου μέχρι τον Φεβρουάριο, τις 19 Φεβρουαρίου. Ναι, 19 Φεβρουαρίου. Παρακαλώ λοιπόν την κυρία Γιαννάκου να αναπτύξει το θέμα της και να μας μιλήσει για την έκθεσή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πολύ σωστά είπατε προηγουμένως ότι η Γιούρη θα κάνει μια απλή γνωμοδότηση και επομένως ε, μαζί της να καθυστερήσουμε κατά ένα μήνα την έγκριση της έκθεσης ούτως ώστε εν τω μεταξύ να υπάρχει και η μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ε, είναι κύριο στοιχείο της δημοκρατικής ζωής μέσα στην Ένωση τα περισσότερα συντάγματα της ένωσης περιλαμβάνουν το ρόλο των κομμάτων μέσα στη δημοκρατική ζωή. Ο σχεδιασμός ενός πακέτου αναδιαμόρφωσης της λειτουργίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των άμεσα συνδεδεμένων με αυτά πολιτικών ιδρυμάτων έχει ως σκοπό πρώτον να διευκολύνει την εσωτερική λειτουργία των ευρωπαϊκών κομμάτων και αφετέρου να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών ώστε να υπάρξει ε, μια πρακτική και άμεση συμμετοχή τους σε αυτά. Τελικός σκοπός είναι η αμεσότερη, μεγαλύτερη και περισσότερη έκφραση των πολιτών στο δημόσιο βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλωσόρισε την πρόταση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σεύκοβιτς η οποία ήρθε σε συνέχεια της έκθεσης ε, της οποίας ήμουν εισηγήτρια το 2011. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι με την έκθεσή μου και το νέο κανονισμό δεν ζητείτε περισσότερη χρηματοδότηση για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αλλά η αναγνώριση ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος τέτοιου που θα επιτρέψει ε, στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να έχουν νομική μορφή αρμόζουσα και όχι αυτή που έχουν σήμερα, δηλαδή μιας διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις τροπολογίες που έχω καταθέσει κύριοι συνάδελφοι, τα σημεία στα οποία υπάρχει κάποιο είδους τροποποίηση είναι, σύμφωνα με τις προτινόμενες τροπολογίες καταρχήν του ε, ε, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Πρώτον είναι τα κριτήρια αναγνώρισης ενός κόμματος ως ευρωπαϊκού. Και πιο ξεκάθαρα, ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα πρέπει να εκπροσωπείται στο 1 τέταρτο των κρατών μελών, δηλαδή τουλάχιστον σε 7 χώρες, από ήδη υπάρχοντα κόμματα, τα οποία έχουν εκλεγμένους βουλευτές στα εθνικά κοινοβούλια ή ευρωβουλευτές τα περιφερειακά κόμματα για να μπορούν να συμμετάσχουν στο σχηματισμό ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος πρέπει να προέρχονται από περιφέρειες στις οποίες αποδίδονται νομοθετικές αρμοδιότητες διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές χώρες υπάρχουν περιφέρειες χωρίς νομοθετικές αρμοδιότητες. Σε κάθε περίπτωση τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να αποτελούν αποτέλεσμα δημοκρατικών διεργασιών και να διέπονται και από τις δημοκρατικές αρχές της Ένωσης. Για να πάρει χρηματοδότηση ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν ευρωβουλευτή. Στην εσωτερική διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος αλλά και στην κατάρτιση των εκλογικών ληστών προτείνω να προωθείτε και να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη η ισότητα των φύλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαπιστώνει ετησίως ότι τα εγγεγραμμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά του ιδρύματα πληρούν όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο registry του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αμφισβητήσει πλήρως δικαιολογημένα σε οποιαδήποτε στιγμή τα κριτήρια εγγραφής ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτείνω η αρμόδια για το θέμα αυτό να αποφασίζει η Επιτροπή να είναι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ή η όποια επιτροπή θα ασχολείται με τα συνταγματικά ζητήματα η οποία μέσα σε δύο μήνες από το αίτημα της επανεξέτασης των κριτηρίων εγγραφής των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα δίνει τη γνώμη της και θα μπορεί να διοργανώσει και ακροάσεις σχετικά με το θέμα. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά του ιδρύματα με τη θέση σε ισχύ του κανονισμού θα έχουν νομική οντότητα η οποία θα αναγνωρίζεται απευθείας υπό την έννοια ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα τελούν υπό το δίκαιο της Ένωσης στην ένομη τάξη του κάθε κράτους μέλους. Θα μπορούν επίσης να μοιράζονται το 90% της χρηματοδότησής τους ανάλογα με το μέγεθος τον αριθμό των ευρωβουλευτών που διαθέτουν ενώ το 10% θα είναι για όλα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα εξίσου. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα θα μπορούν να συμμετέχουν σε δημοψηφίσματα μόνο για θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία της. Και βεβαίως για το κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα θα αναγνωρίζεται μόνο ένα ίδρυμα ως επίσημο και εξαρτώμενο από αυτά. Επίσης τα κόμματα θα μπορούν να υποστηρίζουν ε, εξατομικευμένες καμπάνιες μελών βουλευτών τους ή μελών εθνικών κομμάτων τους μόνο για θέματα που άπτονται των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κύριε Πρόεδρε, η πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προέρχεται βέβαια από δική μας πρωτοβουλία και έγκριση της Επιτροπής μας, ε, έχει τεράστια σημασία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω για τους πολίτες της Ευρώπης. Υπό την έννοια πρώτον ε, ότι κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί ένα πλαίσιο με ευρωπαϊκό χαρακτήρα που δίνει και τη διάσταση της δημοκρατικότητας που πρέπει να έχουν και τα εθνικά πολιτικά κόμματα. Ε, δεύτερον, κατά κάποιο τρόπο νομιμοποιεί ακόμη περισσότερο τη χρηματοδότηση η οποία ήδη υπάρχει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτον, τα κόμματα αυτά τίθενται κατά κάποιο τρόπο όταν χρειαστεί υπό, την, τον έλεγχο κατά κάποιο τρόπο του Κοινοβουλίου εάν αμφισβητηθεί η δημοκρατικότητά τους και η συνάφειά τους με τις ευρωπαϊκές ε, δημοκρατικές αρχές. Και τέλος βέβαια αυτό που έχει ε, νομίζω ιδιαίτερη σημασία είναι ότι αποκτούν συγκεκριμένη βαρύτητα ως πολιτικοί οργανισμοί μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και επομένως να έχουν το ίδιο καθεστώς σε όποιο μέλος, ε, κράτος μέλος και αν εγκατασταθούν το οποίο θα είναι το νομικό καθεστώς που προβλέπεται από τα ευρωπαϊκά όργανα όπως θα αποφασιστεί με βάση το στάτους το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και βέβαια ε, αποτελεί και νομίζω μια σοβαρή προσπάθεια για να γίνει σαφές προς τα έξω ότι αυτό που έχει σημασία και ενδιαφέρει είναι η δημοκρατική τάξη, η καλύτερη σχέση με τους πολίτες της Ευρώπης, γιατί και όλες οι πρωτοβουλίες που η Επιτροπή μας στις οποίες είχε εκπονήσει έκθεση όπως η πρωτοβουλία των πολιτών κτλ. Σε αυτό κατατείνουν, δηλαδή να μπορούν οι πολίτες της Ευρώπης και να γνωρίζουν ποιος κάνει τι και για ποιο λόγο και να έχουν πληροφόρηση. Και ε, να τονίσω κύριε Πρόεδρε τελειώνοντας ότι με την πρόταση της Επιτροπής αλλά και με τη δική μου έκθεση δεν ζητούνται σε καμία περίπτωση περισσότερα χρήματα για τα πολιτικά κόμματα. Για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση ή καμία χρησιμοποίηση αυτής της προσπάθειας η οποία γίνεται ότι δήθεν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή μας ή οι εισηγητές ζητούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Καμία μεγαλύτερη χρηματοδότηση, απλά να δημιουργηθεί η δημοκρατική και ένωμη τάξη που είναι αναγκαία. Σας ευχαριστώ κύριε Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκερέρο έτσι ώστε να αναφερθεί στο δικό του ε, τμήμα, στο τμήμα για το οποίο είναι ε, αρμόδιος. Φαντάζομαι δεν έχουμε ακόμα το έγγραφο της ε, Επιτροπής. Ε, φαντάζομαι ότι θα, φαντάζομαι λέω ότι θα σταλεί και στον, ε, στο, στην Επιτροπή Προπολογισμών. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που ο κύριος Γερέρο έχει ήδη μία έκθεση, νομίζω ότι θα ασχοληθεί καλύτερα με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως, όπως μόλις είπε η κυρία Γιαννάκου, το καθεστώς είναι πρόταση για το νομικό καθεστώς που θα διέπει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τη χρηματοδότησή τους είναι ένα ποιοτικό άλμα πλέον προς τα εμπρός που απορρέει και από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα από την ίδια της την έκθεση της κυρίας Γιαννάκου κατά τη διάρκεια της παρούσης ε, θητείας. Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο δύο λόγια εισαγωγικά θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που θα πρέπει να αποδώσουμε εμείς ε, σε αυτό το θέμα. Να αναγνωριστεί κάτι που ήδη αναγορίζουν οι συνθήκες στο άρθρο 10, αλλά και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο άρθρο 12. Σε αυτά τα δύο άρθρα ορίζεται ότι τα πολιτικά κόμματα τα ευρωπαϊκά εννοώ, συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της κοινή γνώμης και στην έκφραση της πολιτικής βόλησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι ένας παράγον ολοκλήρωσης της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πολιτικά κόμματα είναι θεσμοί που σχηματίζονται από ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά ε, διαδραματίζουν πολύ σημαντικές θεσμικές λειτουργίες. Είναι δηλαδή θεσμοί που με δύο σκέλη. Από τη μια είναι ριζωμένα στην κοινωνία των πολιτών, στην κοινωνία, ε, στην ιδιωτική σφαίρα αν θέλετε, από την άλλη όμως πατούν στο κανονιστικό πλαίσιο των θεσμικών οργάνων και είναι θεσμοί τα κόμματα. Ακριβώς λοιπόν επειδή έχουν ε, θεσμικό ρόλο να διαδραματίσουν θα πρέπει να προστατεύονται από ένα σύστημα που να ρυθμίζει ειδικά το καθεστώς τους και τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που θα πρέπει να έχουν για να ασκούν αυτό το ρόλο που τους αναλογεί, που είναι επαναλαμβάνω ο ρόλος πολιτικής ολοκλήρωσης. Χρηματοδότηση λοιπόν που μας απασχολεί δεν είναι αποκλειστική. Υπάρχουν χώρες και εθνικές ρυθμίσεις που προβλέπουν αποκλειστικά και μόνο δημόσια χρηματοδότηση. Αυτό όμως δεν ισχύει εδώ. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο χρηματοδότησης ιδιωτικής πλέον. Αλλά θα ήθελα να πω και να υπερασπιστώ ότι το γεγονός μόνο ότι υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση είναι ένας παράγον μη διάκρισης που επιτρέπει και εκείνα τα κόμματα που είναι λιγότερο ίσως ελκυστικά για τους ιδιώτες δωρητές να μπορούν να έχουν μια δημόσια στήριξη για να μπορούν να ασκούν ε, τα καθήκοντά τους. Και ταυτόχρονα είναι και ένα κίνητρο καταπολέμησης της παράνομης χρηματοδότησης και τελικά της διαφθοράς. Με άλλα λόγια, η δημόσια χρηματοδότηση εξασφαλίζει. Δεν είναι ένας παράγον που εξισώνει τις δυνατότητες ή τις ευκαιρίες της πολιτικής δράσης των κομμάτων, αλλά σε μεγάλο βαθμό προστατεύει από τις διακρίσεις και προστατεύει και από κάποια παράτυπη χρηματοδότηση ή παράνομη. Για το λόγο αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω της εκθέσεως κυρίας Γιαννάκου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων είναι κατάλληλη και σωστή. Η δική μου τώρα γνώμη, πώς να το πω, πρόταση, όπως είπε και ο Πρόεδρος, αυτή τη στιγμή βασίζεται σε δύο παραμέτρους. Αφενός, δεν υπάρχει επίσημα ακόμα κείμενο που να έχει αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο. Θα το πράξει σε επόμενες ημέρες. Αλλά παρόλα αυτά γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πρότασης αυτής. Χωρίς κείμενο μπορούμε ήδη να εργαστούμε σαν να το είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σαν να είχε αποστείλει επισήμως την πρότασή τη. Ταυτόχρονα όμως δεν είναι προκαθορισμένο ποια θα είναι η καθήλυνα αρμόδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή, ούτε ποια θα γνωμοδοτήσει. Αλλά ε, υποθέτουμε εμείς ότι η καθήλυνα αρμόδια επί της ουσίας θα είναι η Επιτροπή Προεπολογισμών και εμείς θα γνωμοδοτούμε από την ΑΦΚΟ. Πάντως αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούν να ιδωθούν ξεχωριστά. Θα πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού και η ΑΦΚΟ και η ΛΥΜΠΕ. Όπως είπε ο Πρόεδρος, η ΛΥΜΠΕ τελικά δεν θέλει να είναι συναρμόδια επιτροπή ε, με την ΑΦΚΟ επί ίσης αλλά ζήτησε να έχει μια σχέση πιο στενή από τη η σχέση που διέπει τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει ε, αυτό το θέμα τη γνωμοδότηση στη ΛΥΜΠΕ, αλλά τους πρότεινα να μας βοηθήσουν για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα από τα προβλήματα που έχουμε εδώ στον κανονισμό που είναι η συμβατότητα μεταξύ του ευρωπαϊκού δικαίου, ε, του δικαίου των κρατών μελών και του δικαίου της χώρας που έχει την έδρα του ε, κάθε πολιτικό κόμμα, κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Είναι τρεις ένοπες τάξεις λοιπόν, ευρωπαϊκή, εθνική και η χώρα στην οποία δράβει το κόμμα. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη συνεργασία, μεγάλο συντονισμός για να μην αντιμετωπίσουμε νομικά ε, προβλήματα έτσι κάποιες εμβέλειας. Εγώ επικεντρώνομαι στο θέμα που μου αναλογεί, όπως είπε και η κυρία Γιαννάκου ήδη, η δική της έκθεση, η πρόταση για το νέο καθεστώς δεν περιλαμβάνει δημοσιονομικές υποχρεώσεις νέες. Δηλαδή, δεν ζητάει περισσότερα χρήματα. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο αλλάζει ο κανονισμός χωρίς να αυξάνεται η χρηματοδότηση. Ε, αλλάζοντας όμως ο κανονισμός και το καθεστώς, έχουμε μια νέα απέτηση Υπάρχουν κάποιοι γενικοί δημοσιονομικοί κανόνες τη Ένωση, στους οποίους θα πρέπει να εγγράφεται και αυτή η πρόταση, χωρίς, επαναλαμβάνω, να αυξάνεται η χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει να ενταχθεί εδώ ένα νέο κεφάλαιο που να αναφέρεται ειδικά στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά του ιδρύματα, διότι, όπω σα είπα και προηγουμένω, και στην έκθεση της κυρίας Γιαννάκου τα λέει αυτά. Έχει γίνει μια αναθεώρηση τώρα του τρόπου χρηματοδότησης και των κομμάτων αλλά και των ιδρυμάτων. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσω κάτι ακόμα. Εδώ στην Επιτροπή μας, σε προηγούμενες συνεδριάσεις, ανέκαθεν προτείναμε να έχουμε πιο σαφείς κανόνες για τα πολιτικά κόμματα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο συστηματικά ζητούσαμε ένα καθεστώς με τη στενή έννοια για τα κόμματα αυτά και να ε, υπάρχει και κατάλληλη χρηματοδότηση. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τόσο το καθεστώς όσο και η πρόταση αναθεώρησης των οικονομικών κανόνων ανταποκρίνονται σε αυτή μας τη δέσμευση. Επίσης, στο παρελθόν η έκθεση της κυρίας Γιαννάκου και το Κοινοβούλιο ζητούσε κάποιες αλλαγές. Και αλλάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το σύστημα που ίσχυε με δωρεές, grants, και τώρα το ονομάζει συνεισφορές, contributions. Βεβαίως υπάρχει διαφορά. ανάμεσα στη χρηματοδότηση των κομμάτων και των ιδρυμάτων. Νομίζω ότι είναι προφανές. Υπάρχουν και αντικειμενικές διαφορές ανάμεσα σε ένα πολιτικό κόμμα και ένα ίδρυμα πολιτικό. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αλλά επίσης θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι σε πολλές στιγμές του δημοκρατικού γίγνεσθε τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα ε, έχουν κοινούς στόχους και κοινέ στρατηγικές μακροπρόθεσμα. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι καλό να γίνει τόσο αυστηρός διαχωρισμό ανάμεσα στη χρηματοδότηση των κομμάτων και των ιδρυμάτων. Απόλυτα υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερότητε. Εντάξει, άλλο το κόμμα, άλλο το ίδρυμα, αλλά δεν θα πρέπει να είναι αεροστεγής αυτή η ε, χρηματοδότηση. δεν είναι τελείως διαφορετικές οντότητες. Πολύ συχνά συνεργάζονται και έχουν τους ίδιους στόχους και την ίδια στρατηγική και το ίδιο πεδίο λειτουργίας. Δεν θα μπω τώρα στο καθεστώς, τα είπε η κυρία Γιαννάκου. Προβλέπει αυτό τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να σέβονται ε, τις βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης και τη μη διάκριση και τους κανόνες εσωτερικής δημοκρατίας και τη διαφάνεια. Αυτά είναι αρχές βέβαια, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται και για τη χρηματοδότηση. Τα κόμματα θα πρέπει να είναι διαφανή, να λογοδοτούν για τη χρηματοδότησή τους και να εξηγούν Πώς γίνεται η διαχείριση των πόρων που θα τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο λεπτομερή και λογιστικό. Δηλαδή, να γίνονται σεβαστές αυτές οι αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και στις δαπάνες, αλλά και να υπάρχει και μια αναλογικότητα. Δηλαδή, τους δίνουν κάποιους πόρους για κάποιο σκοπό. Σε αυτό το σκοπό θα πρέπει να δαπανώνται οι πόροι αυτοί. Αλλά δεν θα πρέπει να δημιουργούμε άχρηστα εμπόδια στην ομαλή λειτουργία των κομμάτων για να μην τα κάνουμε γραφειοκρατικά μορφώματα ε, υπερβολικά άκαμπτα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρηματοδότηση αυτή καθ' αυτή ως εισηγητής, αναγνωρίζω ότι έχει νόημα να υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο στους δημοσιονομικούς κανόνες και θα φέρει τον τίτλο Συνεισφορέ στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα» μέσα στους κανόνες δηλαδή τους οικονομικούς της Ένωσης νομίζω ότι είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που να αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αυτό από μόνο του τους δίνει μια αξία, μια ειδική αναγνώριση και ενισχύει αυτό που σας είπα προηγουμένως το θεσμικό ρόλο τελικά που ε, παίζουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Επίσης, θεωρώ θετικά κάποια άλλα στοιχεία έτσι πιο λειτουργικά. Δηλαδή, καταργείται η χρηματοδότηση γύρω από ένα ετήσιο πρόγραμμα και τελικά θα είναι μία χρηματοδότηση για λειτουργία των κομμάτων που εκ των υστέρων θα πρέπει να έρχονται να τη δικαιολογούν. Δηλαδή, δεν θα είναι πάντα συνδεδεμένη η χρηματοδότηση με την κατάθεση ενός προγράμματος εκ των προτέρων θα παίρνουν κάποια χρήματα για τις δραστηριότητές τους τις οποίες όμως θα πρέπει να δικαιολογούν και ως προς την εκτέλεση των ε, κονδυλίων αυτών. Και αυτό θετικό είναι. Μπορεί να γίνει και κάποια μεταφορά από ένα χρόνο στον άλλο όταν υπάρχει ένα απόθεμα στον προπολογισμό ή κάποια συγκεκριμένη δυνατότητα για ένα ποσό και για μια περιορισμένη χρονική διάρκεια να μπορεί να μεταφέρεται από το ένα χρόνο στο άλλο και να είναι, θέλετε, έτσι μια προκαταβολή της δραστηριότητας του κόμματος για το επόμενο έτος. Βεβαίως είμαι υπέρ και νομίζω όλοι μας εδώ στην Επιτροπή μας να υπάρχει και έλεγχος αλλά και κυρώσεις εκ των υστέρων και πάλι αυστηρές που να δείχνουν ότι τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι υποδειγματικά στη λειτουργία τους. Τίποτα δεν καταστρέφει περισσότερο την αξιοπιστία των ε, πολιτικών κομμάτων και των θεσμών στα μάτια της κοινή γνώμης από την έλλειψη των ελέγχων ή από τις πλημελείς ελέγχους ή από τις αμφιβολίες ε, κατά πόσο έχουν δαπανηθεί σωστά κάποιοι πόροι από τα θεσμικά όργανα ή από τα κόμματα. Ή όταν θεωρούν οι πολίτες ότι όλα αυτά συμβαίνουν με αδιαφάνεια ή ότι συγκαλύπτονται και υπάρχει ατιμορρησία σε περίπτωση ατασταλιών. Θα πρέπει λοιπόν και οι κυρώσει και η τιμωρία να είναι παραδειγματική και αυστηρή. Όταν αποδεικνύονται αντικανονικές συμπεριφορές ως προς τη χρηματοδότηση. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει εδώ στην Επιτροπή μας, που είναι το εξής. Τι γίνεται με τις προεκλογικές εκστρατείες. Εδώ δεν ε, προβλέπεται ένα ειδικό καθεστώς χρηματοδότηση εν ώψη εκλογών. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τουλάχιστον την ε, χρονιά που προηγείται των ευρωεκλογών, έχουν αυξημένη δραστηριότητα από την κανονική τους λειτουργία. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να δεχθούμε ότι εντάξει δεν υπάρχει δική χρηματοδότηση για την προεκλογική εκστρατεία, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το προηγούμενο έτος πριν τις εκλογές ενδεχομένως η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα του κόμματος, δηλαδή να είναι αυξημένη σε σχέση με την κανονική του χρηματοδότηση. Τελειώνω. Αν θυμάστε την πρόταση που ήταν ακόμα άτυπη, ανεπίσημη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει μια σειρά σημείων εκεί στοιχείων που αναφέρονται οι αλλαγές για τη χρηματοδότηση. Και πρέπει να σας πω, και θα κλείσω εδώ, ότι εμείς, εγώ δηλαδή καταρχήν ως εισηγητής της έκθεσης ή της νομοδότησης, ε, συμφωνώ να καταργηθεί η χρηματοδότηση βάσει ετησίου προγράμματος εργασιών, γιατί έτσι είναι μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του κόμματος και της δραστηριότητάς του. Δεν υπάρχει αυτό σε κανένα κράτος μέλος να καταθέτει ένα πρόγραμμα εργασιών, ένα κόμμα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων βάσει πραγματικών δαπανών και όχι βάσει χρηματοδότησης κάποιων δράσεων που έχουν προγραμματιστεί και στο μέλλον ενδεχομένω να υλοποιηθούν. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Και όπως προτείναμε και εμείς να είναι ξεκάθαρη η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην επιλεξιμότητα ενός πολιτικού κόμματος σε σχέση με τα κριτήρια που ισχύουν για να εγγραφεί αυτό το κόμμα και να δηλωθεί και να αναγνωριστεί ως Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. Είπα ότι συμφωνώ να αυξηθεί η δυνατότητα αποθεματικού καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς για μια διετία των απορρόφητων κονδυλίων και όπως προτείνει και η κυρία Γιαννάκου θεωρώ ότι είναι καλό να μειωθεί ο συντελεστής συγχρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, γιατί έτσι αν μειωθεί αυτό, τα λιγότερο ισχυρά ας πούμε, κόμματα μπορούν ουσιαστικά να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία και με μεγαλύτερη αυτονομία. Και τέλος, το γεγονός ότι ενισχύονται οι κυρώσεις, ότι υπάρχει ένα καθεστώς ελέγχου από πλευράς της Όλαφ και του Ελεκτικού συνεδρίου ε, είναι ευπρόσδεκτες προτάσεις. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει και αυτό ρόλο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της λειτουργίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Και στο ως προς το σεβασμό των αρχών. Δεν λέω να έχουν την ίδια θεώρηση για την Ευρώπη, ούτε το ίδιο όραμα, ούτε να θεωρούν την Ευρώπη ως πολιτικό γίγνεσθε. Δεν μπορούν να αποκλείονται με αυτά τα κριτήρια κάποια κόμματα. Μπορεί κάλλιστα να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που να έχει ως στόχο την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που να μην τηρεί τους δημοκρατικούς κανόνες που ισχύουν γενικώ και από την έννοια αυτή λοιπόν στηρίζω την πρόταση και της κυρίας Γιαννάκου. Δηλαδή μία από τις αρχές αυτές θα πρέπει να είναι η μη διάκριση για... Και τέλος, και τελειώνω όπως είπαμε, θα προσπαθήσω μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το ποια θα είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και ποια θα γνωμοδοτήσει, επειδή θα έχουμε και στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου την επόμενη συνεδρίαση, Μέχρι τότε θα φροντίσω, αλλιώς για το Γενάρη, να σας φέρω ε, και τροπολογίες. Γιατί μόλις μάθαμε ότι μέχρι το Φεβρουάριο δεν πρόκειται να ψηφίσουμε αυτές τις δύο εκθέσεις. Και της κυρίας Γεννακού και τη... Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν παρεμβάσεις ε, επί αυτών των δύο ε, παρουσιάσεων, εκθέσεων. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί εγγεγραμμένοι. Ho già dato la parola al collega Egnio. Έδωσε το λόγο, έδωσε ήδη το λόγο στον συνάδελφο Άγνιου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν είμαι πολύ γνωστός εδώ στην Επιτροπή σας, γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μιλήσω πρώτος. Λοιπόν, εγώ είμαι Ευρωβουλευτής για άνω των τριών ετών και ξέρω ότι εδώ στο κάμπους των Βρυξελών βλέπει κανείς όλο καινούργια κτίρια και δίνεται η εντύπωση ότι κυκλοφορούν σημαντικοί άνθρωποι και άρα όλα καλά τα κάνει το κοινοβούλιο. Αλλά τι λένε οι εκλογείς. Δεν είναι πολύ εντυπωσιασμένοι γιατί όλο και λιγότεροι ψηφίζουν στις ευρωεκλογέ. Αυτό τους λέει το ένστικτό τους και στη χώρα μου το Ηνωμένο Βεσίλειο όχι μόνο έχει μειωθεί η συμμετοχή στις ευρωεκλογέ, αλλά και οι λίγοι αυτοί που ψηφίζουν ψηφίζουν όλο και περισσότερο με, για το UKIP που είναι κατά της συμμετοχής στην Ένωση. Άρα στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει πολύ λίγη υποστήριξη προς το όργανο αυτό. Και άρα δεν υπάρχει μία πραγματική εντολή για τη δημιουργία πανενωσιακών κομμάτων. Πού είναι η εντολή. Κόμματα που ανακαλυπτουν και τις 27 χώρες μέλη λέει τι λένε οι ψηφοφόροι μας. Ψηφίζουν όλο και λιγότεροι, αλλά πολύ περισσότεροι στις εθνικές τους εκλογές, γιατί ξέρουν ότι εκεί βρίσκεται η εξουσία και εκεί θέλουν να βρίσκεται. Δύο πράγματα με ανησυχούν. Το ένα είναι τα χρήματα και το άλλο τα δημοψηφίσματα. Για τα χρήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθαρός εισφορέας, δίνει πάρα πολλά λεφτά και δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση κομμάτων που μπορεί στη Βρετανία να μην γίνουν ποτέ αποδεκτά ε, εξτρεμιστικές οργανώσεις που τις χρηματοδοτούμε εμείς. Δεν μας αρέσει αυτό. Μια στιγμή. Και το άλλο θέμα που δεν μου αρέσει είναι ότι αυτή η ιδέα της χρηματοδότησης των φορολογουμένων εμείς οι φορολογούμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρηματοδοτούμε κανένα κόμμα. Γιατί να το κάνουμε στην Ευρώπη για τα δημοψηφίσματα τώρα, για ενωσιακά θέματα. Αυτό είναι θέμα των χωρών. Και τα λεγόμενα πανενωσιακά κόμματα δεν δικαιολογούνται καθόλου να διοργανώνουν δημοψηφίσματα. Τώρα για την ισορροπία των φύλων εδώ πρόκειται για προσβολή προς τις εκλογές. Υπάρχουν περισσότερες γυναίκες μεταξύ των εκλογέων από το όσο άντρες γιατί ζουν περισσότερο. Αλλά δεν προσφεύγουν, δεν καταφεύγουν τις εκλογές για να ψηφίσουν γυναίκες, άντρες ψηφίζουν. Και δεν τους λέμε όχι, δεν ισχύει αυτό πρέπει να είναι περισσότερες γυναίκες, όχι πρέπει να ακούμε τη φωνή του εκλογέα ό,τι και να μας πει. Μπορεί να το θεωρείτε εσείς άνηση μεταχείριση. Προσφύγετε στα δικαστήριά σας, πλάκα θα έχει. Αλλά μέχρι πού θα πάνε όλα αυτά. Μήπως και το ομοφιλόφιλο περιεχόμενο της κοινωνίας πρέπει να εκπροσωπείται αναλογικά ή οι κοκκινομάλιδες ή οι γαλαζομάτιδες Πού θα σταματήσει αυτό το γλίστριμα. Σεβαστείτε επιτέλους τι λένε οι εκλογείς. Και τέλος, τι θα γίνει τελικά σε αυτές τις εκλογές. Βλέπετε ότι η κρίση του ευρώ στην Ελλάδα και αλλού δείχνει, ε, δημιουργεί άνοδο των εξτρεμιστικών κομμάτων και αυτά θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο και στις ευρωεκλογές θα εμφανιστούν και όλα αυτά δεν είναι καθόλου υγιή και σας ζητώ όλους να βγείτε από εκεί μέσα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αγνίου. Ο κύριος Νταφ. Κοιτάξτε. Καλησπέρα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι εκτός από εκείνους βέβαια που δεν το θέλουν που δεν αναγνωρίζουν τις πολιτικές πραγματικότητες δηλαδή, ότι τα πανενωσιακά ευρωπαϊκά κόμματα θα γίνουν κάτι όλο και σημαντικότερο γιατί προσπαθούν να οικοδομήσουν μια βιώσιμη και όρημη υπερεθνική δημοκρατία. Και το ψήφισμά μας του Στρασβούργου της περασμένης Πέμπτης, ε, παρεμπιπτόντως ευχαριστώ όσους το υποστήριξαν. Το ψήφισμα λοιπόν εκείνο που ζητάει από τα πολιτικά κόμματα να ορίσουν τους υποψηφίους τους και το πρόγραμμά τους για τις επόμενες ευρωεκλογές αποτελεί ένα ποιοτικό άλμα προς την σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα δε να ευχαριστήσω την κυρία Γιαννάκου και τον κύριο Γκερέρο για την παρουσίαση που έκαναν των σκέψεών τους και των αντιδράσεών τους προς τις προτάσεις της Κομισιόν. Διαβάζοντάς τες κι εγώ, τις βρίσκω πιο τεχνοκρατικές από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά αν η Κομισιόν πραγματικά καταλαβαίνει ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης των πολιτικών κομμάτων. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλά λεπτά προβλήματα που θα συζητηθούν στον τριμερή διάλογο και δεν βλέπω να γίνεται σύντομη συμφωνία με βάση τις προτάσεις αυτές. Ιδιαίτερα ανησυχητικό για μένα είναι το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να εγγράφονται στα κράτη. Πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει τρομερές ανομαλίες. Ανάλογα βέβαια με την κατάσταση του κάθε κόμματος και βεβαίως θα καταλήξει σε άνηση μεταχείριση κατά της πλήρους χρηματοδότησης των, της προεκλογικής εκστρατείας των πανενοσιακών ή ομοσπονδιακών κομμάτων. Νομίζω ότι η Κομισιόν, πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να δημιουργήσει πέρα από τα υπόλοιπα και έναν καθεστώς για τις ε, οργανώσεις που δεν είναι κερδοσκοπικές, ιδιαίτερα δε για τα ομοσπονδιακά πολιτικά κόμματα. Πράγμα το οποίο θα έκανε τα πράγματα σαφέστερα και πιο ισότιμα. Με βάση το οποίο να κάνουν την καμπάνια τους τα κόμματα αυτά. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να πούμε κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω για τον δημοκρατικό ρόλο τους, διότι δεν είναι αποδεκτό να χρηματοδοτούμε πολιτικά κόμματα αν επιβάλλονται όλες οι αποφάσεις από τον πρόεδρό τους. Πρέπει να επιμείνουμε για τη δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων που χρηματοδοτούνται, για διαφάνεια και δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έγκριση του καθεστώτος, του καταστατικού των πολιτικών κομμάτων, του προγράμματός τους, τον ορισμό των αξιωματούχων τους και ίσως και την επιλογή των υποψηφίων τους. Μιλάω πάντοτε για τις διεθνικές λίστες και ψηφοδέλτια. Βέβαια μόλις το 14 θα ισχύσουν όλα αυτά, αλλά πρέπει από τώρα να τα οργανώσουμε. Τρίτον, θα ήθελα να επιμείνω στην άδεια που πρέπει να έχουν αυτά τα ενωσιακά πολιτικά κόμματα να συμμετέχουν σε εθνικά δημοψηφίσματα για ευρωπαϊκά θέματα. Θα ήταν παράλογο να απαγορεύσουμε την συμμετοχή τους εφόσον είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκού χαρακτήρα κόμματα άρα έχουν άμεσο συμφέρον και ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Αυτά είναι τα τρία σημαντικότερα σημεία και αντιρρήσεις που έχω μέχρι τώρα και προσβλέπω σε στενότερη συνεργασία με τους δύο συνεισηγητές για να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση εδώ μέσα. ώστε να καταλήξουμε στην διαπραγματευτική εντολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Φόξ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα δεν ξέρω αν ο συνάδελφος θέλει να τελειώσει το τηλεφώνημά του, μπορεί να πάει και έξω από την αίθουσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία που έκανε για την έκθεση αυτή. Ε, δεν έχω τίποτα εναντίον των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων όντως εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της Ευρώπης μακάρι να ήθελαν ε, να ε, συμμετέχουν σε αυτό το, σε αυτό το ε, τη διαδικασία και αυτό θα δείξει ότι είναι μια νίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εδώ βλέπουμε ότι τα κόμματα αυτά στηρίζονται από τα χρήματα των φορολογουμένων. Εγώ όμως δεν συμφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι ε, νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε τα κοινά ευρωπαϊκά χρήματα έτσι ώστε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήθελαν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχει βεβαίως ε, κάποια ευθυγράμμιση μεταξύ των ε, πολιτικών κομμάτων και όταν κάποιος θέλει να μπει σε μια πολιτική ομάδα λαμβάνει υπόψη του κυρίως τις πολιτικές συνάφειες και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και να το λάβουμε υπόψη μας. Ο κύριος Γκερέρο λέει ότι δεν θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα αλλά θα αλλάξει ο τρόπος ε, κατανομής. Αυτό όμως ε, σημαίνει ότι τα, περισσότερα χρήματα θα πάνε στα μεγαλύτερα κόμματα και τα λιγότερα στα μικρότερα κόμματα. Φαντάζομαι ότι δεν εκπλήσωμε που στα μεγάλα κόμματα είναι το ΕΛΚ και το, ε, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό όμως να υπάρχουν εδώ απαιτήσεις απέτηση δηλαδή ότι το ε, κόμμα αυτό θα πρέπει να ε, εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο γιατί ενδεχομένως θα υπάρξει με τον τρόπο αυτό διακριτική μεταχείριση έναντι κάποιων άλλων πολιτικών ε, σχηματισμών. Δεν θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια ότι το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε εθνικά δημοψηφίσματα. Και σας εξηγώ γιατί. Γιατί και στις 27 χώρες έχουμε διαφορετικές νομοθεσίες και θα έχουμε διαφορετικές νομοθεσίε ε, που θα σχετίζονται και με το τι μπορεί να γίνει ή τι δεν μπορεί να γίνει ε, ε, πάντα σε αναφορά με το σύνταγμα της κάθε χώρας. Επομένως, το να επιβάλλουμε ένα κανονισμό που να λέει ότι ανεξάρτητα του τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο αυτά τα χρήματα θα πρέπει να πηγαίνουν στην εκστρατεία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα κυρίως δε στις μικρότερες χώρες όπου μπορεί το αποτέλεσμα να είναι δυσανάλογο ε, της χρήσης αυτών των χρημάτων. Εάν οι εθνικές νομοθεσίες επιτρέπουν τέτοιου είδους δαπάνες, ναι, ε, θα μπορούσαν ε, τα κόμματα να διαλέξουν να ξοδέψουν τα χρήματά τους με τον τρόπο που θέλουν. Αλλά νομίζω ότι στις μικρές χώρες ε, εάν αυτά τα τεράστια κόμματα του ΕΛΚ ή του, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχουν μια τεράστια δύναμη πυρός, τότε θα μπορέσουν να αλλάξουν υπέρ τους την ψήφο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η οδός είναι ολιστηρή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δεν είμαι υπέρ της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων είτε από τον Εθνικό Προϋπολογισμό είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιούνται άσχημα τα δημόσια χρήματα δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, αλλά μπορεί να γίνει και χειρότερο. Ε, εάν ε, τα κόμματα αυτά τελικά ε, αποφασίσουν ε, να, συν, να συνεργάζονται έτσι ώστε να δημιουργήσουν και, και κάποιες αρχές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν υποχρεωτικά και τα άλλα πολιτικά κόμματα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο και ακόμα χειρότερη χρήση του δημοσίου χρήματος. Το θέμα βέβαια είναι και όλα ποιοι θα είναι είναι υποψήφοι για τα κόμματα αυτά και ε, με τι είδους ε, προϋποθέσεις ε, θα μπαίνουν αυτοί οι υποψήφοι. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ δημοκρατικά όλα αυτά αυτή ε, η χρήση της ε, ε, δημοκρατίας και που χρησιμοποιείται έτσι λίγο σαν μπαχαρικό για να φτιάξει τη γεύση οτιδήποτε λέμε ή κάνουμε δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης μακροπρόθεσμα το κατά με απασχολεί το κατά πόσον θα περάσουμε σε μια κατάσταση όπου τα πολιτικά, ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα είναι σε θέση να κερδίσουν ευρωπαϊκές εκλογές και ξέρετε ε, καμιά φορά το δυνατό γίνεται πιθανό, έτσι γίνεται. Ε, εδώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χέφνερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σα ευχαριστώ πολύ εσά κύριε Γιαννάκου και κύριε Γκερέρο Σαλόμ για την τόσο καλή προετοιμασία των εκθέσεων. Από τη φύση των πραγμάτων της συζήτησης ε, αυτής στην Επιτροπή θα αναγκαστώ να περιοριστώ ε, σε κάποια ζητήματα που χρειάζονται συζήτηση. Δεν θα επαναλάβω τα επιτυχημένα ή τα λιμένα ζητήματα. Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα ή να πω ε, τι θα ήθελα να ξανασυζητήσουμε. Και αρχίζω από αυτό που θεωρώ σημαντικότερο. Και είναι ενδιαφέρον που το συζητούσαμε κάθε φορά αυτό το θέμα και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει εδώ μια σαφή τάση στην Επιτροπή μας, τουλάχιστον στο παρελθόν, στην ακρόαση που κάναμε πέρσι, όλοι οι εμπειρογνώμονες, χωρίς καμία ε, εξαίρεση, είπαν ότι είναι μεγαλύτερη αδυναμία και θα πρέπει να αλλάξει επιγόντως. Αλλά δεν βλέπω ουσιαστική ακόμα απάντηση στο εξή ερώτημα στην έκθεση. Και το ερώτημα είναι Μα να το πω αλλιώς, είναι μια αναγκαιότητα. Η εγγραφή, η καταχώρηση των πολιτικών κομμάτων, πώς είναι δυνατόν να διαχωρίζεται από τη χρηματοδότηση. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ε, είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια. Άλλο είναι η χρηματοδότηση. Στη χρηματοδότηση θα πρέπει να έχουμε και κάποια κριτήρια επιτυχίας. Δηλαδή, το θεωρώ θεμητό να χρηματοδοτούνται ανάλογα με την επιτυχία τους τα κόμματα. Δηλαδή, όταν έχουν περισσότερες ψήφους, να είναι και μεγαλύτερη η χρηματοδότησή τους, γιατί έχουν μεγαλύτερη απήχηση στο λαό. Αυτοί που έχουν μικρότερη απήχηση στο λαό να παίρνουν μικρότερα, λιγότερα χρήματα και να υπάρχει και ένα κατόφλι. Και όταν κάποιο κόμμα κινείται κάτω από το κατόφλι αυτό, να μην τίθεται θέμα αποζημίωσης. Τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά ως προς την καταχώρηση, την εγγραφή του κόμματος. Η εγγραφή θα πρέπει να πληρεί κάποια τυπικά κριτήρια, όχι κριτήρια επιτυχίας. Ας πούμε, αν έχει επαρκή οργάνωση, αν έχει πρόγραμμα, αν έχει καταστατικό, αν έχει μέλη, ε, ταχύ μέλη, δεν ξέρω κάποιον αριθμό μελών, να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις και τυπικές και ουσιαστικές, ανεξαρτήτως αριθμού ψηφοφόρων ας πούμε, για το χάρτη των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων και όλα τα άλλα που συζητήσαμε. Εφόσον πληρούνται αυτά τα κριτήρια, θα πρέπει κατά την άποψή μου ένα κόμμα να μπορεί να καταχωρείται, να επιτρέπεται να εγγράφεται ως Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα όταν πληρεί τα ουσιαστικά αλλά και τα τυπικά προσόντα και τις προϋποθέσεις. Ακόμα και αν δεν το ψηφίσουν αρκετοί ψηφοφόροι για να χρηματοδοτηθεί. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι προ όφελο τη ευρωπαϊκή δημοκρατία και το λέω πολύ συνειδητά και στο δικό μα συμφέρον θα πρέπει να είναι να μην δημιουργούμε ούτε μονοπόλια ούτε ολιγοπόλια κομμάτων. Αλλά όσο γίνεται ένα μεγαλύτερο ο ανταγωνισμό να επιτρέπεται ελευθερία και εδώ να διαγωνίζονται ας πούμε διάφορα πολιτικά κόμματα και ιδέες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να αφήσουμε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κλειστό όμιλο, ας πούμε ένα κλαμπ και να αποκλείουμε κάποιους άλλους που παρόλα αυτά πληρούν τα κριτήρια. Και θέλω να ρωτήσω και την κυρία Γιαννάκου και τον κύριο Γκερέρο, γιατί δεν έχω καταλάβει ακόμα ακριβώς τι γίνεται. Αυτές οι τόσο διαφορετικές αρχές που ισχύουν για τη χρηματοδότηση και για την εγγραφή των κομμάτων. Πώς θα ρυθμιστεί αυτό στην πράξη και πώς θα διατηρηθούν ξεχωριστά αυτά τα δύο. Να πω κάτι ακόμα για τη χρηματοδότηση, μια ακόμα ερώτηση που έχω. Έχει νόημα, πιστεύω, για τη χρηματοδότηση αφενός να υπάρχει ένα κατόφλι, παράδειγμα, να υπάρχει μια στοιχειώδης χρηματοδότηση για τη διατήρηση της οργανωτικής δομή και μετά ανάλογα με την εκλογική επιτυχία. Στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 15% του βασικό και 85% του ποσού εξαρτάται από την επιτυχία του κόμματος. Εσείς θέλετε να τα αλλάξετε, να το κάνετε 10% και 90%. Γιατί? Δεν έχω καταλάβει γιατί το 15-85 το θεωρούσα καλός, ε, τεκμηριωμένο, ε, αιτιολογημένο. Και θα παρακαλούσα να διατηρηθεί, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί το αλλάζετε, γιατί το κάνετε 10 και 90. Και μια άλλη ερώτηση για την τροπολογία υπαριθμών 3 και σε σχέση με τις τροπολογίες 13 με 17, εάν τις είδα καλά. Σε ποιο βαθμό τα πολιτικά κόμματα που τηρούν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα το κρίνουμε εμείς. Αυτό ζητάει η συγκήτρια. Και ρωτώ, η δική μας επιτροπή είναι καλή ιδέα. Εμείς όλοι εδώ εκπροσωπούμε κάποια πολιτικά κόμματα. Εμείς δεν θα ήμασταν καν μέλη του Κοινοβουλίου ούτε της Επιτροπής μας εδώ, εάν δεν ήμασταν σε ψηφοδέλτια πολιτικών κομμάτων και δεν είχαμε εκλεγεί. Και το θεωρώ σχετικά προβληματικό αυτό το θέμα, ειδικά επί της ουσίας, έτσι, για θέματα α, της ουσίας. θα τα κρίνει αυτά. Εμείς τα μέλη τη Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων θα αποφασίζουμε για άλλα κόμματα. Ακόμα και τότε, αν έχουμε αποχρόντες λόγους και κατόπιν ορίμου σκέψεως ε, αποφανθούμε, θα τον αμφισβητήσουν στην κοινή γνώμη τουλάχιστον εκείνοι οι οποίοι θίγονται και πάντα θα μπορούν να μας προσάπτουν ότι θέλουμε να προστατευτούμε από τον ανταγωνισμό, να αποκλείσουμε ανταγωνιστές και άλλα τεινά δεν θα ήταν πολύ πιο ευφιές αυτή την απόφαση να την αναθέσουμε σε ένα ανεξάρτητο όργανο, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και αν αυτό το όργανο που πρέπει λίγο να συζητηθεί, να καταλήξουμε σε ποιο θα είναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα για τη δημοκρατική εσωτερική δομή και διάρθρωση. Έχω λίγο την αίσθηση ίδια με τον Άντριου Νταφ σωστά το προσεγγίζετε, αλλά νομίζω ακόμα δεν είναι αρκετή η ρύθμιση και η διατύπωση. Δηλαδή, Όταν έχουμε εσωτερικές αρχαιρεσίες ε, για τα διοικητικά όργανα, τα προεδρία των πολιτικών κομμάτων ή ακόμα και για κατάλογους ε, υποψηφιολίστες, ψηφοδέλτια, θα πρέπει να υπάρχει μια εσωτερική δημοκρατική δομή και λειτουργία του κόμματος και να είναι προϋπόθεση και για την καταγραφή του κόμματος αλλά και για ε, τη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέπουμε τη λειτουργία ούτε να δίνουμε χώρο σε μη δημοκρατικά κόμματα. Και ποιος αποφασίζει αν είναι δημοκρατικό το κόμμα ή όχι, δεν είναι μόνο η στόχη του, αλλά είναι και η ίδια του η λειτουργία στο εσωτερικό, αν είναι δημοκρατικό το κόμμα. Παράδειγμα, στη Γερμανία χρειάστηκε να επαναληφθεί ολόκληρη εκλογή κάποτε, ε, για το λόγο και μόνο ότι όταν καταρτίστηκαν τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων, ε, το συνέδριο του κόμματος που έκανε το ψηφοδέλτιο, που γι' αυτό το λόγο είχε συγκληθεί, δεν είχε τη δυνατότητα να αποφασίσει για κάθε θέση του ψηφοδελτίου, αλλά το Προεδρείο ε, είχε καταθέσει μια πρόταση, ένα έτοιμο ψηφοδέλτιο που μπορούσε κανείς μόνο κάτω από κοπή να το εγκρίνει, να το απορρίψει. Γι' αυτό και μόνο το λόγο λοιπόν χρειάστηκε να επαναληφθεί ολόκληρη εκλογή στη Γερμανία. Ε, γιατί ήταν παράνομο στη γερμανική τάξη ακριβώς επειδή δεν είχε καταρτιστεί το ψηφοδέλτιο με δημοκρατικά κριτήρια. Τώρα δεν θέλω εγώ να επιβάλλω στην Ευρώπη ούτε να συστήσω το γερμανικό δίκαιο, αλλά νομίζω ότι η δημοκρατική απόφαση για τον τρόπο που καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια, γιατί είναι από τις βασικότερες αποφάσεις που καλείται να λάβει ένα κόμμα, είναι σημαντικό γιατί τα κόμματα, αν θέλετε, στρατολογούν ε, το ανθρώπινο δυναμικό για τα κοινοβούλια. Και ένα από τα κριτήρια θα πρέπει να είναι αυτό, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται δημοκρατικά και η απόφαση αυτή εντός ενό κόμματο. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ. Για το θέμα των δημοψηφισμάτων, αυτή η διάμεση λύση που προτάθηκε, δηλαδή να μην επιτρέπει τη συμμετοχή του σε δημοψηφίσματα εκτός αν πρόκειται για ευρωπαϊκά θέματα, δεν με πείθει πάρα πολύ αυτό το επιχείρημα. Γιατί μετά θα ερχόμαστε να διαπληκτιζόμαστε αυτό το θέμα είναι ευρωπαϊκό ή δεν είναι. Και ποιο δεν είναι ευρωπαϊκό. Ε, θα πρέπει να το ρυθμίσουμε με τη ώρα που πιο σαφή αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να ε, φύγω για λίγο, γι' αυτό λοιπόν ε, παρακαλώ την Αρχολογρήπη να, πάρει, να αναλάβει μάλλον την Προεδρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και νομίζω ότι η συγγήτρια θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι η συγγήτρια και στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και στις 4.30 έπρεπε να είμαι εκεί, έτσι ώστε να παρουσιάσω και εκεί την έκθεσή μου. Το σημειώνουμε. Έχουμε όμως ε, τέσσερις αγορητές που έχουν εγγραφεί, γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, να είναι όσο γίνεται πιο σύντομοι. Ο Σάνθος Βέμπερ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καταρχάς πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι ότι αυτή η πρόταση και η ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημαίνει ένα ποιοτικό άλμα σημαντικό αυτό το θέμα της νομικής μορφής των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, κομμάτων θα πρέπει λέει να ρυθμίζεται με βάση το κράτος το οποίο έχουν την έδρα τους. Αυτό είναι λίγο προβληματικό. Θα πρέπει να σκεφτούμε ίσω ευρωπαϊκέ δομέ εδώ, όχι εθνικέ. δεύτερο, η σύνδεση της ίδρυσης ενό τέτοιου κόμματο με τον αριθμό των βουλευτών, των ερετών και στα εθνικά κοινοβούλια ή τα περιφερειακά, αν έχουν ήδη ερετού, είναι κάτι το θετικό, αλλά έτσι αποκλείουμε την ίδρυση κομμάτων αυθόρμητα από πολίτες. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα κίνημα πολιτών που θέλει να δημιουργήσει Ευρωπαϊκό Κόμμα. Ξέρω εγώ ένα κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης που θέλουν να στοιχηθούν μαζί οι πολίτες και να δημιουργήσουν Ευρωπαϊκό Κόμμα. Δεν μπορούν ε, με την παρούσα πρόταση. Θα πρέπει να έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε κάποιο επίπεδο στη χώρα τους. Εντάξει λοιπόν είναι καλό πρώτο βήμα αλλά για το μέλλον δεν θέλω να αποκλείσω τη δυνατότητα ε, τα κινήματα πολιτών να δημιουργούν Ευρωπαϊκά κόμματα. Ένα τρίτο και αυτό με βασανίζει πολύ και συμφωνώ και έχει δίκιο ο κύριος Χέφνερ για την έγκριση των κομμάτων. Λέει μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόταση. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγγράφεται το κόμμα αυτό στη λίστα και παίρνει την έγκριση. Δηλαδή ποιο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ολομέλεια, έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα στην Ολομέλεια θα αποφασίσουμε εάν ένα κόμμα ε, ακροδεξιό ή ακροαριστερό εγγράφεται ως ευρωπαϊκό. Δεν μπορώ να το φανταστώ πάρα πολύ εύκολο αυτό. Στέλνουμε αποστολές στην Αφρική παρατήρησης εκλογών και η πρώτη ερώτηση που κάνουμε είναι είναι ελεύθερη ίδρυση των κομμάτων ή θα πρέπει να ζητήσουν την άδεια κάπου να καταχωρηθούν σε ένα μητρό. Και θα το κάνουμε αυτό στην Ευρώπη και μάλιστα θα επαφείται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η απόφαση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για την έγκριση, τον έλεγχο των κριτηρίων χρειαζόμαστε ένα όργανο ουδέτερο, ανεξάρτητο και ακριβώς δεν θα πρέπει να είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί στο Κοινοβούλιο συγκρούονται τα κόμματα μεταξύ τους είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό και το τελευταίο για το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών και πάλι θα ζητούσα εδώ κατά την ίδρυση των κομμάτων να αφήνουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο περιθώριο. Τι θα λέγαμε εμείς στο Κοινοβούλιο αν ε, ιδρυόταν ένα αποκλειστικά γυναικείο κόμμα για την ενίσχυση των γυναικείων δικαιωμάτων. Ας πούμε, ε, ορισμένες γυναίκες συγκροτούν ένα κόμμα. Αν βάλουμε κριτήριο φύλου, δεν θα μπορέσει το κόμμα να ιδρυθεί γιατί δεν υπάρχει ισορροπία φύλου. Και εδώ θα παρακαλούσα να υπάρχουν κάποια ελάχιστα κριτήρια, δημοκρατία, κράτος δικαίου, αλλά να μην το παρακάνουμε στα κριτήρια. Ευχαριστώ. Merci. La parole est à notre collègue, Madame Tain. Ευχαριστώ, η συνάδελφος κυρία Τάιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ ρητά να πω ότι θέλω ευρωπαϊκά κόμματα με ένα χωριστό ευρωπαϊκό καθεστώς, όπως είπε και ο συνάδελφος Βέμπερ. Δηλαδή το δικό μας το φιλελεύθερο κόμμα θα πρέπει να ιδρυθεί με βάση το βελγικό δίκαιο. Ε, δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το γνωρίζω το βελγικό δίκαιο και για να είμαι δεν έχω και την όρεξη να καθίσω να ασχοληθώ με 27 ξεχωριστέ νομοθεσίε. Είναι αρκετά δύσκολο να γνωρίζει κανεί την ίδια του την νομοθεσία. Οπότε προτιμώ ευρωπαϊκό. Θα ήθελα να πω στο συνάδελφο Άγνιο που έχει φύγει βέβαια, ότι από τη Γερμανία ε, υπάρχει το συνταγματικό δικαστήριο, δεν θεωρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως γνήσιο κοινοβούλιο και αυθεντικό. Γιατί εγώ έχω εκλογή από Γερμανούς ψηφοφόρους και συναποφασίζω και για τους Βρετανούς. Και αυτό μπορεί να θεωρεί. Θα πρέπει να έχουμε ε, κάποια στιγμή μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ένα ευρωπαϊκό δήμο εντός εισαγωγικών και ε, επίση για τη χρηματοδότηση. Τα είπε και ο συνάδελφο Χέφνερ και με κάλυψε. Ε, θα πρέπει να σας πω ότι ακριβώς εκεί που είναι μεγάλο το κόστος, παράδειγμα, σε ένα συνέδριο κόμματο, που είναι αρκετά ακριβή διοργάνωση, στο συνέδριο του κόμματο των φιλελευθέρων, σε διεθνές επίπεδο, ευρωπαϊκό δηλαδή, έρχονται λιγότεροι βουλευτές συνεδροί από ότι ε, ένα συνέδριο των φιλελευθέρων στη Γερμανία. Οπότε η σημασία των ευρωπαϊκών κομμάτων δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Ε, δεν συμφωνώ πάρα πολύ για τα ιδρύματα. Έχουμε μεγάλη νομολογία στη Γερμανία. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ίδρυμα και το κόμμα μπορεί και τα δύο να συνεισφέρουν ε, στη διαμόρφωση της κοινή γνώμης πολιτικά, αλλά είναι πολύ μεγάλες διαφορές. Και στη χρηματοδότηση χρειάζεται τεράστια προσοχή. Και όντως να υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα ιδρύματα. Για τις κυρώσεις τώρα, ε, και τα κόμματα. Εγώ δεν περιμένω πάρα πολλά από τις κυρώσεις. Βλέπω να, να αποθέτεται μεγάλες προσδοκίες στην Όλαφ και τα λοιπά. Εντάξει, παίζει ρόλο η Όλαφ, αλλά οι αποφάσεις της δεν είναι δεσμευτικές. Και αν κοιτάξετε κάνει το ελεγκτικό συνέδριο, την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ψηφίσαμε τον προπολογισμό και είχαμε μία παράγραφο που έλεγε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για 16η φορά ε, θεωρεί απαράδεκτο τον προπολογισμό, δηλαδή θεωρεί ότι δεν μπορεί να απορροφηθεί αυτό ο προπολογισμό και αυτή η παράγραφο αφαιρέθηκε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, ο έλεγχο χρειάζεται εκ των προτέρων, πιστεύω εγώ, και εκ των υστέρων. Και για τη διαδικασία έγκριση ενό κόμματο, βέβαια δεν μπορεί καμιά επιτροπή, ούτε η δική μα εδώ, ούτε κανεί άλλο να ελέγχει επί τη ουσία το περιεχόμενο του κόμματο, ούτε κάνει ολομέλεια. Αυτό αντιτίθεται στη διάκριση των εξουσιών, για να το πω έτσι. Μόνο ένα δικαστήριο μπορεί να αποφαίνεται, όχι κοινοβούλιο. Κάποιο ανεξάρτητο σώμα, όργανο, δεν ξέρω ε, με ποια σύνθεση. Πάντω όχι βουλευτές, καλά ποτέ δεν είναι 100% ανεξάρτητο ένα όργανο. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε ποια είναι η τελευταία ε, δομή που θα αποφασίσει. Ο συνάδελφος ανέφερε προηγουμένως το κόμμα των γυναικών. Ε, λέμε ότι θα εγκρίνονται κόμματα που δεν θα εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών. Στο κόμμα μου ε, κάναμε μια ψηφοφορία σε εθνικό επίπεδο και δεν ξέρω κατά πόσο το δικό μου κόμμα θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στην Ευρώπη. Μάλλον δεν θα τις πληρούσε με τη σημερινή του δομή. Ε, κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Και ε, σε ό,τι αφορά τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, χρηματοδοτούμε πολλέ. Ε, που προπαγανδίζουν αντιευρωπαϊκά θέματα και μας ε, υπονομεύουν. Νομίζω και αυτό ανήκει στη δημοκρατία. Δηλαδή, το σύνορο ποιο είναι. Η συνταγματικότητα και μόνο. Όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να επιτρέπονται. Δηλαδή και όλοι οι Βρετανοί, όλα τα κόμματα που είναι κατά της Ευρώπης θα πρέπει να ε, επιτρέπονται. Τι θα γίνει, θα απαγορεύσουμε τώρα τα Βρετανικά κόμματα που είναι ευρωσκεπτιστικά στην Ολομέλεια. καταψηφίσαμε και διάφορα ε, άλλα θέματα που στις χώρες μας μπορεί να ισχύουν και για τον κύριο Νταφ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μπορούν, επιτρέπεται τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να συμμετέχουν. Μα πώς θα γίνει διαφορετικά. Τα κόμματα αυτά έχουν την καλύτερη γνώση, πραγματογνωμοσύνη, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Δεν ξέρω, τυπικά ή άτυπα. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σεφλίνγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οθήθηκα να απαντήσω από τους κυρίους Φόξ και Άγνιου για τα δημοψηφίσματα μου φαίνεται ότι δημοψήφισμα για ευρωπαϊκό θέμα σε μια χώρα μέλος επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες. Η ίδια η Ένωση δηλαδή είναι ενδιαφερόμενος στην περίπτωση αυτή. Όσο για τη συμμετοχή στις εκλογές, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει σε κάθε δημοκρατία μία τάση για χαμηλότερη συμμετοχή στις εκλογές, για περισσότερη αποχή. Και αυτό επηρεάζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια και οφείλεται κυρίως στην αύξηση άλλων σωμάτων με πολιτική εξουσία μεταξύ των οποίων και θέσεις στην κοινωνία των πολιτών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ένωσης. Τώρα, πιθανές κυρώσεις πρέπει να καθορίζονται με αντικειμενικό τρόπο και διαδικαστικά και ουσιαστικά και να είναι διαφανέστατες έπειτα. Το θέμα εισόδου-εξόδου από το σύστημα. Εδώ χρειάζεται μια αποσαφήνιση. Η ένταξη πρέπει να είναι ανοιχτή αλλά όχι απόλυτη. Από την άλλη, ζούμε σε καιρούς αρκετά ασαφής και μερικές οργανώσεις μπορεί να θέλουν να μπουν σε κάποιο πολιτικό σύστημα για λόγους ε, δευτερεύοντες για να μην πω τριτεύοντες. Παραδείγματος χάρη σε πολλές χώρες, εγώ σκεφτόμαι τρεις, υπήρξαν κόμματα με πολύ περίεργους τίτλους τα οποία έζησαν πάρα πολύ λίγο. Και αυτό μπορεί να ισχύσει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Τελευταίος ο μιλητής κύριος Ήλτσεφ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος γιατί η κυρία Γιαννάκου πρέπει να φύγει έτσι ώστε να παρουσιάσει την έκθεσή της στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να της ευχηθούμε θάρρος και επιτυχία στην ε, εργασία της ε, γιατί προκύπτουν πολλά ζητήματα στη συζήτηση αυτού του θέματος. Και γιατί. Όχι, γιατί όχι μόνο προσπαθούμε να ε, εισάγουμε κάτι καινούριο, όχι μόνο θέλουμε να ξαναδούμε από άλλη σκοπιά ε, το ε, ευρωπαϊκό έτσι, πολιτικό σύστημα, αυτό που σχετίζεται με τα κόμματα τουλάχιστον, αλλά θέλουμε και να βρούμε απαντήσεις σε νέα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Ας πούμε συμμετοχή μεγάλο των μεγάλων κομμάτων στις μικρές χώρες η ιδέα είναι βεβαίως ότι εάν μεγάλα κόμματα με πολλά χρήματα έρθουν σε μικρές χώρες ε, ενδεχομένως θα καταστρέψουν τις, ε, τα μικρότερα κόμματα. Ε, αυτό συνέβη λίγο και τη δεκαετία του 90 όταν έγιναν οι πολύ μεγάλες αλλαγές και είδαμε ότι όταν ας πούμε άνοιξαν μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων πολυεθνικών κτλ καταστράφηκαν τα μικρά μαγαζιά, κυρίως στις μικρές πόλεις. Ε, νομίζω πάντως ότι οι μικρές αυτές χώρες χρειάζονται ε, και ευρωπαϊκή εμπειρία, όχι για οτιδήποτε άλλο, τουλάχιστον για να σταματήσει ας πούμε η πολιτική χειραγώργηση. Ε, η Βουλγαρία είναι μια μικρή χώρα, έχουμε 200 ε, καταχωρισμένα κόμματα και επομένως ακολουθώντας και την λογική μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα καλό επιτυχές αποτέλεσμα έτσι ώστε ε, να ε, γίνει και πιο σαφές το πολιτικό τοπίο σε πολλές χώρες. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να οφαλοσκοπούμε, να σταματήσουμε αυτές τις εγωκεντρικές θέσεις, να πούμε ότι χρειαζόμαστε την στήριξη κάποιων πολιτικών ε, ομάδων ή κάποιων πολιτικών οικογενειών. τώρα υπάρχουν κόμματα κόμματα βεβαίως πιο μεγάλα όπως το ΕΛΚ, όπως οι φιλελεύθεροι που περιμένουν ότι θα εκλέξουν μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών ε, ε, και βεβαίως αναμένεται οι υπόλοιποι να πρέπει να κάνουν κάποιο συμβιβασμό. Νομίζω ότι εάν στην έκθεση ε, προβληθεί αρκετή διαφάνεια τότε αυτοί οι συμβιβασμοί θα είναι μικρότεροι θα είναι λιγότεροι. Ε, θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις. Ε, νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, εάν δηλαδή οι προϋποθέσεις είναι σωστές. Όσον αφορά τώρα τα δημοψηφίσματα, αυτά θα πρέπει να γίνουν με συμμετοχή μεγάλη. Ας πούμε, στις 27 Ιανουαρίου στη χώρα μου το, το, του 2013 θα γίνει δημοψήφισμα για την ε, πυρηνική ε, ενέργεια. Ε, ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι νοσταλγοί της Σοβιετικής Ένωσης και θα ψηφίσουν με έναν τρόπο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν πιο ευρωπαϊκό προσανατολισμό θα ψηφίσουν διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εάν κρατήσουμε δημιουργήσουμε ε, μία βασική χρηματοδότηση ε, και εάν αμβληθεί αυτή η ιδέα ότι κλέβονται κατά κάποιο τρόπο τα ευρωπαϊκά χρήματα όλα θα είναι καλύτερα. Δεν νομίζω ότι ε, ότι ο Ευρωπαίος ε, ε, ψηφοφόρος ε, θα είναι απογοητευμένος και δεν θα θελήσει να ψηφίσει για τέτοια κόμματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Η συγγήτρια κυρία Γιαννάκου θέλει σύντομα να σχολιάσει. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Κυρία Πρόεδρε μου σύντομα. Ε, εγώ ξεκαθάρισα από την αρχή ότι δεν τίθεται θέμα αύξηση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν. Εκπλήσωμαι με ορισμένους συναδέλφους που κάνουν σαν να έγιναν σήμερα τα πολιτικά κόμματα. Τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν και χρηματοδοτούνται. Δεύτερον, είναι άλλη η καταχώρηση ενός κόμματος και άλλη η χρηματοδότηση δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αν δεν έχει τουλάχιστον ένα ευρωβουλευτή. Τρίτον, το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει πολιτικές απόψεις, αλλά το Κοινοβούλιο είναι που χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό του. Και το Κοινοβούλιο οφείλει να ελέγξει αν ένα κόμμα ανταποκρίνεται στις αρχές και τις αξίες της Ένωσης και στις δημοκρατικές αρχές. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι επειδή το Κοινοβούλιο είναι πολιτικός οργανισμός όλοι είναι μία αντικειμενικοί αυτό δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο θέμα. Στα δημοψηφίσματα φυσικά και μπορούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αφού μπορούν τώρα που δεν έχουν νομική μορφή, δεν θα μπορούν να τα αναποκτήσουν. Αυτά είναι περίεργα που ακούω. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι γιατί φοβάμαι ότι υπάρχει σύγχυση. Τα πολιτικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα αποκτήσουν αυτή τη νομική μορφή η οποία θα αναγνωρίζεται έτσι κι αλλιώς από όλα τα κράτη-μέλη. Θα υπερισχύει η νομική μορφή του κανονισμού. Δεν θα είναι σε κάθε κράτος μέλος ό,τι θέλει όποιος θέλει. Και είναι δικαίωμα ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος και τότε και τώρα και τώρα να εγκατασταθεί όπου του αρέσει. Το ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι στις Βρυξέλλες δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάνε στη Μαδρίτη ή στην Αθήνα ή όπου θέλουν Δηλαδή μην παριστάνουμε σαν να μην το ξέρουμε το θέμα, σαν να μην υπάρχουν πολιτικά κόμματα και έρχονται τώρα για πρώτη φορά ξαφνικά. Τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν και χρηματοδοτούνται. Και επαναλαμβάνω δεν είναι θέμα ούτε να πάρει χρήματα κάποιος από κάποιον άλλον, ούτε να αυξηθούν τα χρήματα. Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται ένας κανονισμός ή μία οδηγία και αποτελεί υποχρεωτικά δίκαιο για τα κράτη μέλη με τον ίδιο τρόπο θα αποτελεί και αυτός ο κανονισμός δίκαιο για τα κράτη μέλη και δεν έχει λόγο να έρχεται σε αντίθεση εφόσον θα είναι κάτω από τις δημοκρατικές αρχές της ένωσης με το καθεστώς που υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος εκτός αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν κράτη μέλη που έχουν μη δημοκρατικές αρχές για τα κόμματά τους οπότε τότε είναι ένα ερωτηματικό τι γίνεται στα κράτη μέλη αλλά δεν είναι ώρα να μπούμε σε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ήθελα από τους συναδέλφους προτάσεις ή ζητήματα που θέλουν να ξεκαθαρίσουν σε σχέση με την έκθεση ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε με διαβούλευση ε, και συνεννόηση γιατί αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά σε όλους μας. Δεν αφορά μόνο ε, σε μία πλευρά και βεβαίως για τα ιδρύματα δεν μπορεί ένα κόμμα να έχει δέκα ιδρύματα ούτε μπορεί ένα κόμμα να έχει κοινοβουλευτική ομάδα μία στο ευρωκοινοβούλιο και πέντε κόμματα απ' έξω. αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. δηλαδή δεν θα φτιάξουμε κάτι που θα το μεταχειρίζονται ορισμένοι κατά το δοκούν. επομένως οι κανόνες θα είναι κανόνες. αν θέλει ένα κόμμα να αναγνωρίζεται ως ευρωπαϊκό και επομένως να έχει και το αντίστοιχο κύρος και να μην είναι μη κυβερνητική οργάνωση όπως είναι σήμερα στο Βέλγιο εγώ νομίζω ότι ούτε νομικά θέματα ανακύπτουν, ούτε προβλήματα θα υπάρξουν. Θα υπάρχουν πέντε κριτήρια για να αναγνωρίζετε το κόμμα, κριτήριο για να χρηματοδοτείτε το κόμμα, δυνατότητα των πολιτών να αμφισβητούν το κόμμα και βεβαίως εάν θέλετε να προσθέσουμε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια τριμελή επιτροπή από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να ελέγξει αν ένα κόμμα είναι δημοκρατικό, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ότι πιο αναλυτικά και πιο σωστά θα εξήταζε το θέμα η Επιτροπή που ασχολείται με τις ε, θεσμικές υποθέσεις. Επομένως δεν υπάρχει αντίρρηση σε σχέση με αυτό. Αλλά ο προβληματισμός που εξετέθη από ορισμένου συναδέλφους με εξέπληξε. Γιατί είναι σαν να μην έχουμε ξανασυζητήσει για τα κόμματα και σαν να μην υπάρχουν κόμματα. Μα τα κόμματα υπάρχουν. Παίρνουν χρήματα από το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν κόμματα που έχουν πάρει χρήματα από το Κοινοβούλιο χωρίς να δικαιούνται. Λοιπόν, μην ε, εμφανιζόμαστε τώρα και λέμε ξαφνικά ότι τι γίνεται και πώς θα γίνει με την έκθεση. Αν κοιτάξετε τις προηγούμενες εκθέσεις θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν δεν, δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνα. Είναι γνωστά όλα αυτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία εισηγήτρια, κυρία Γιαννάκου. Ε, νομίζω ότι διευκρινίσατε πολλά πράγματα ε, και τώρα νομίζω ότι ο κύριος Γκερέρο θα θέλει να μιλήσει και αυτό για το δημοσιονομικό κανονισμό. Ευχαριστώ. Μετά από αυτή την παρέμβαση της κυρίας Γιαννάκου, έτσι με τόσο πάθος και συμφωνώ με στο πνεύμα της, ήθελα να πω ότι επειδή προέρχομαι από μια χώρα ε, έτσι καθολική στην παράδοσή της και με ένα παρελθόν που συνδέεται πάρα πολύ με την αντιμεταρρύθμιση τη Συνόδου του Τρέντο. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι εστί μανιχαϊσμός. Δηλαδή, δημιουργείς κάτι που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα και πας να το πολεμήσεις. Και πολλά από αυτά που ακούσαμε είναι μανιχαϊστικό. Δηλαδή ότι πάμε να πολεμήσουμε κάτι που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Πουθενά εδώ δεν λέει ότι θα οριστεί με ποιο τρόπο κάθε κόμμα επιλέγει την ε, διεύθυνσή του ή τα διοικητικά του όργανα. Γενικά με δημοκρατικούς τρόπους. Πουθενά δεν λέει ότι τα πολιτικά ε, κόμματα θα πρέπει να ε, συμβουλεύονται το εκλογικό τους πρόγραμμα. Όταν μπαίνουμε στα συγκεκριμένα ζητήματα, τότε θα απαντήσουμε και να απαντήσω στις μερικά συγκεκριμένα που ακούσαμε. Υπάρχουν δύο-τρία ζητήματα κλειδιά. Το είπε ο κύριος Χέφνερ και είναι η κλασική συζήτηση που γίνεται εδώ στην Επιτροπή μας. Να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στα προαπαιτούμενα για να αναγνωριστεί ένα πολιτικό κόμμα, να εγγραφεί ως Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα και ε, τα προπετούμενα και τα κριτήρια για να χρηματοδοτείται ως Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. Για το πρώτο, για την αναγνώριση, είναι αντικειμενικά τα κριτήρια. Και δεν ε, έχουν καμία σχέση με πολιτικό πρόγραμμα. Καμία όμως. Το είπα στην αρχή, αν θέλει ένα πολιτικό κόμμα να ιδρυθεί για να καταπολεμά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ε, πλήρως ε, εναρμονισμένο με τον ισχύοντα κανονισμό. Αλλά ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που να προτείνει να γίνονται διακρίσεις για λόγους θρησκείας, για λόγους κοινωνικής τάξης, φιλής ή φίλου, δεν ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το μόνο που πρέπει να κάνει το Μητρό των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων είναι να διαπιστώνει ότι δεν παραβιάζονται οι βασικές πολιτικές ε, αρχές. Από την άλλη πλευρά είναι τελείως διαφορετικό το ζήτημα της χρηματοδότησης. Εκεί χρειάζεται απλούστατα το κόμμα αυτό να έχει μια κάποια απήχηση στο λαό. Αλλιώ δεν θα υπήρχε καμιά διαφορά ανάμεσα στη χρηματοδότηση ενό κόμματο που αντιπροσωπεύει 30% των Ευρωπαίων και ένα άλλο που εκπροσωπεί 2.000 ευρωπαίου πολίτε. Και εδώ τώρα μπορεί κανεί να μπει σε μια συζήτηση, όπω έκανε ο κύριο Χέφνερ, αν είναι 10 και 90, 85, 15, χρηματοδότηση και τα ποσοστά. Το λογικό είναι να υπάρχει μια σημαντική χρηματοδότηση που να συνδέεται με τον ε, την απήχηση εν πάση περιπτώσει που έχει το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα στα μάτια του λαού. Και όποια και να είναι η πρόταση αυτή, 10, 90, 85, 15, θα είναι πάντα με φθήνουσα αναλογικότητα. Δηλαδή, τα μικρά κόμματα τελικά θα είναι ευνοημένα από αυτή τη ρυθμίση, σε σύγκριση αναλογικά πάλι με τα μεγάλα. Κάτι άλλο που είπαν πολλοί, ο κύριος Νταφ, ο κύριος Χέφνερ, διευκρίνηση την νομική μορφή που θα έχει ε, το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση έτσι ώστε να μην συζητάμε συνεχώς εάν ισχύει το βελγικό δίκαιο ή κάθε κράτος μέλους ή αν ισχύει το ίδιο το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ποια είναι η νομική μορφή. Αυτό θα πρέπει να το λύσουμε κάποια ώρα. Με τρόπο σωστό. Ένα τρίτο σημαντικό ζήτημα που συζητήθηκε και αυτό είναι ποιο είναι το όργανο τελικά που απορρίπτει ένα ε, πολιτικό κόμμα. Είτε ε, διότι ε, το καταστατικό του δεν συνάδει με τις βασικές δημοκρατικές αρχές της Ευρώπης, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε διότι έχει μια συμπεριφορά που αντιφάσκει με το καταστατικό. Δεν ασκεί σωστά τη λειτουργία και τα δικαιώματα. Λοιπόν, ποιος το ορίζει αυτό. Τώρα μπορεί ο καθένας να προτείνει διάφορα. Έχει νόημα η αντίσταση αυτή που υπάρχει να μην είναι μόνο το κοινοβούλιο, υπάρχει μια προστασία δικαστική τελικά, μια δικαιοδοτική σε τελική φάση. Να μην αποφασίζει μόνο το κοινοβούλιο. Το κοιτάξουμε, αυτό θέλει δουλειά ακόμα. Ένα τελευταίο που θέλω να σας πω τώρα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπλέξω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί μπορεί να είναι έτσι σχετικά συγκρουσιακό, αλλά το λέω με την κάθε ε, προσωπική φιλία και προσύνια. Εδώ η Επιτροπή μας κυριαρχείται ε, αντιπροσωπεύονται οι Βρετανοί και καμιά φορά και οι Γερμανοί. Ε, επειδή εδώ επικυριαρχούν λοιπόν οι Βρετανοί, ε, δίνουν την εντύπωση ότι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μια και από την άλλη ο κόσμο όλο. Είναι πολύ σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι μία από τις 27 χώρες της Ένωσης, όσο σημαντική και να είναι. Και πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να λυθούν στο εσωτερικό του, εν πάση περιπτώσει. Και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν κατά ανάγκη ε, όλα τα ζητήματα που αποφασίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, εάν θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει δημοψήφισμα για το αν ανήκει ή όχι στην Ένωση, με γεια του, με χαρά του. Δεν πρόκειται κανείς να το εμποδίσει, να το κάνει το δημοψήφισμα. Αλλά έχει δικαίωμα. Όπως έχουν και άλλες χώρες. Αυτό γιατί θα πρέπει να επηρεάσει το σύνολο της νομοθεσίας στην Ένωση. Και όταν λέω ότι υπερεκπροσωπείται και η Γερμανία, είναι με διαφορετική μορφή εναγκαλίζονται συνεχώς ε, την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαστηρίου για να επιχειρηματολογούν. Ωραία. Το άκουσα αυτό και δεν το λέω για πρώτη φορά. Α, ξέρετε γιατί εγώ εκλέγομαι στη Γερμανία αλλά παίρνω αποφάσεις που επηρεάζουν τους Βρετανούς. Ωραία. Και αυτό εδώ πέρα το μαγαζί λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, με τον ίδιο τρόπο ένας βουλευτής που εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια της Ματρίτης παίρνει αποφάσεις που αφορούν εξίσου ε, τους βουλευτές και τους πολίτες που ζουν στη Βαρκελόνη και στη Σεβίλη. Λοιπόν, είτε είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν είμαστε. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο γερμανικός λαός λέει έχει μια ειδική ξεχωριστή ταυτότητα τόσο ιδιαίτερη που μόνο όταν γίνονται σεβαστές αυτές οι ιδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο τότε θεωρείται δημοκρατικό. Δημοκρατικό είναι ότι την χή ημέρα του 2014 εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίων θα ψηφίσουν για τις ευρωεκλογέ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι εκπρόσωπος των πολιτών, των Ευρωπαίων, όλων. Και με τον ίδιο τρόπο που είπα προηγουμένως για τους Βρετανούς, και οι Γερμανοί θα πρέπει να το λύσουν στο εσωτερικό της Γερμανίας τη σχέση τους που έχουν με το συνταγματικό τους δικαστήριο. Δεν ξέρω αν επεκτάθηκα ή αν παραφέρθηκα, <laughs> αλλά Εντάξει, ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να τα πω, εν πάση περιπτώσει αυτά. Merci. Ε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Βλέπουμε ότι η μελέτη αυτών των ε, ε, εκθέσεων μας οδηγεί σε πολύ πυκνές πολιτικές, σε πολύ συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα. Ναι, ε, θα έχω ένα διαδικαστικό. Θα τα πω περίπου ισπανικά, ισπανοπορτογαλικά. Να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ο μανιχαϊσμός δεν έχει καμία σχέση με τη μεταρρύθμιση, ε, με την αντιμεταρρύθμιση και ε, με τη σύνοδο του Τρέντου. Ο μανιχαϊσμός είναι μια φιλοσοφία ε, του τρίτου αιώνα μετά Χριστόν που το εφήβρε ο Αυγουστίνος και μετά το κατέριψε και ο Αυγουστίνος. Αυτό το ενδοϊσπανικό καθολικό πρόβλημα που είναι ένα θέμα του εμφυλίου πολέμου της Ισπανίας το έχει ξεπεράσει η, ανθρωπότητα. Ναι, εγώ λέγομαι Ρίκη Αυγουστίν, λέει Αυγουστίνος. Γιατί είναι και 28 Αυγούστου η γιορτή του Αγίου Αυγουστίνου, μεγάλη χάρη του. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για αυτήν ε, την ε, ε, υψηλή έτσι, ανταλλαγή πολιτικών και ιστορικών απόψεων. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε όλα τα έγγραφα μεταφρασμένα ε, για την επόμενη συνεδρίασή μας 17-18 ε, Δεκεμβρίου. Στις 19 Ιανουαρίου θα κάνουμε την τελευταία συζήτηση και στις, 19 Φεβρουαρίου, στις 20 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε στην, έκθεση, στην ε, Επιτροπή μας. Τώρα, βάσει της ημερησίας διατάξεως προβλέπεται κοινή συζήτηση επί δύο εκθέσεων. Η πρώτη έκθεση αφορά την τροποποίηση του κανονισμού που ε, σχετίζεται με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρχής Ε, όσον αφορά ε, τα νέα καθήκοντα, ειδικά καθήκοντα για την προληπτική εποπτεία των πιστοτικών ιδρυμάτων και μετά έχουμε μία έκθεση επί της οποίας πρέπει να συντάξουμε γνωμοδότηση και αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν πάλι την προληπτική εποπτεία των πιστοτικών ιδρυμάτων. Ε, για την πρώτη έκθεση η είναι ο κύριος Παύλο Ραγγέλ, για την δεύτερη ο κύριος Άντριου Ντάφ είχαμε ήδη την δυνατότητα στην τελευταία μα έκτακτη συνεδρία στου Στρασβούργο την εβδομάδα να ακούσουμε του δύο εισηγητέ. Δεν ξέρω εάν τώρα οι εισηγητέ έχουν παρατηρήσει ή σχόλια επιπλέον ε, κυρίω όσον αφορά τι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί από τα μέλη της Επιτροπής μας. Ο κύριος ε, ε, Ραγγέλ μήπως θέλει να πάρει το λόγο έτσι ώστε να μπορέσει να σχολιάσει ίσως κάποιες από τις ε, τροπολογίες του. Ναι. Νομίζω, λέει ο κύριος Ραντζέλ, ότι δεν υπάρχει λόγος ε, να αναφερθώ σε βάθος ε, στις τροπολογίες αυτές. Συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι πιο παραγωγικό και καλό θα ήταν να ακούσουμε τα σχόλια των συναδέλφων, εάν και εφόσον έχουν τέτοια σχόλια. Και βεβαίως μετά πρέπει να πω ότι θα είμαι απολύτως στη διάθεση των συναδέλφων να απαντήσω στα διάφορα ερωτήματα ή σχόλια τα οποία θα έχουν καταθέσει. Ο κύριος Ντάφ όμως μήπως θέλει να πάρει το λόγο, ναι. Έχετε τώρα τις τροπολογίες, το έγγραφο με τις τροπολογίες και βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές συμβαστικές ε, τροπολογίες ε, οι οποίες ε, προέκυψαν βάσει των σχολείων που έκαναν διάφοροι συνάδελφοι και πολιτικές ομάδες. εκτός από την ΚΟΕ. Ε, διότι ο κύριος Σόλτς ε, έχει επιλέξει μια εναλλακτική οδό την οποία σέβομαι μεν αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ ρεαλιστική. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό δηλαδή τώρα να θεωρήσουμε ότι ε, θα ε, να δημιουργήσουμε τώρα μία ενιαία αρχή η οποία θα προκύψει από την σύνθεση τις ρυθμιστικές αρχές τις οποίες έχουμε ε, καθορίσει ήδη το 2010. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάντως θα βρίσκεται ούτως ή άλλως στον ε, πυρήνα, ε, θα βρισκόταν στον πυρήνα της ενιαίας εποπτικής ε, αρχής. Βεβαίως μπορούμε να κρατήσουμε την ιδέα μελλοντικής σύγκλησης των μεμονωμένων ρυθμιστικών αρχών ε, μετά το πέρας μιας πρώτης αναθεωρητικής περίοδου ενδεχομένως. Πάντως είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να προχωρήσει έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι τοποθετήσεις του, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες χώρες μέλη οι οποίες προσπαθούν λίγο να αποσταδρομήσουν σε σχέση με τις αρχικές θέσεις που είχαν ε, ε, πάρει στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό. Δηλαδή, εάν αποτύχουμε, εάν δεν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την οικοδόμηση της ε, Τραπεζικής Ένωσης όσο γίνεται πιο γρήγορα, τότε τα μηνύματα τα οποία θα στείλουμε προς τα έξω, προς τις αγορές και προς τους ψηφοφόρους θα είναι καταστροφικά. Όπως ξέρετε έχω προσπαθήσει να αναφέρω ότι τα ε, ε, ζητήματα αυτά θα πρέπει, ε, συγγνώμη, ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν την αρχή και να έχουν ίδια δικαιώματα, ε, δηλαδή η Ευρωζώνη και η μη Ευρωζώνη ε, να έχουν τα ίδια ε, δικαιώματα. Είναι τέτοια η φύση των συμβατικών υποχρεώσεων και έτσι ώστε να είναι σαφές ότι οι κεντρικές τράπεζες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Επίσης, ότι η εποπτική αρχή ε, θα πρέπει να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω άμεσων προτάσεων, ε, δηλαδή προσχέδια αποφάσεων. Ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δια του Διοικητικού της Συμβουλίου θα πρέπει ε, να μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει ε, βάσει ε, ενισχυμένης πλειοψηφίας αυτές τις προτάσεις. Επίσης, αναφέρω μία διαδικασία για την εκλογή της, του Εποπτικού Συμβουλίου. που βέβαια βάζει η διαδικασία αυτή το Κοινοβούλιο σε μια πολύ ισχυρή θέση. Θα ήθελα να ακούσω σχόλια από τους συναδέλφους όσον αφορά ε, τις συμβαστικές ε, τροπολογίες που προτείνω. Αναλογιζόμενος ε, την συζήτηση που είχαμε στο Στρασβούργο, νομίζω ότι μέσω των τροπολογιών προσπάθησα να ενσωματώσω και τις ε, απόψεις των άλλων πολιτικών ομάδων. Να προχωρήσουμε λοιπόν έτσι ώστε να φτάσει το θέμα και στην Επιτροπή ε, ε, ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Γκερέρο πρώτα. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι όμως πάρα πολύ σύντομος διότι η τοποθέτηση μου αφορά την έκθεση του κυρίου Ρανζέλ που έχει 10 τροπολογίε. Πέντε είναι δικέ μου. Και μου έστειλε και συμβιβαστικές, τι οποίες δέχομαι. Σε σχέση με την έκθεση αυτή, είναι σημαντικό το θέμα της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, να υπάρχει ένας έλεγχος πιο τυποποιημένος και άλλα ζητήματα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν παρεμβάσεις περισσότερο επί της ουσίας για την έκθεση του κυρίου Νταφ, αλλά δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκουαλτιέρη είχε επίσης ζητήσει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. ένα πολύ ειδικό θέμα σε σχέση με το συμβασμό προτείνει ο Έντριου. Σε γενικές γραμμές στηρίζω την έκθεση. Αναφέρομαι όμως στο συμβιβασμό C. Στην ΕΚΟΝ έχει επιτευχθεί επίσης μια καλή συμφωνία όσον αφορά τον ε, ορισμό του ε, επικεφαλής του Προέδρου μάλλον ε, της Συμβουλευτικής Αρχής και είπαμε διασυνενέσεως του Κοινοβουλίου αναρωτιέμαι μήπως θα ήταν πιο ρεαλιστικό και λαμβάνοντα υπόψη και την συμφωνία που έχει επιτευχθεί στην ΕΚΟΝ, μήπως ε, να ε, ακολουθήσουμε ακριβώ την ίδια διαδικασία. Ε, maybe slightly more Νομίζω ότι να πούμε, αντί να, να πούμε ας πούμε ότι είναι appointed by the parliament, και ενδεχομένως εδώ να έχουμε τη δυνατότητα για ε, προφορική τροπολογία αυτής της συμβαστική τροπολογίας. Ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι μήπως ζητούν το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένως θα ζητήσω από τους δύο εισηγητές να απαντήσουν. Παροραγγέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και στη δικιά μου έκθεση έχουμε τη γραμμή Γκουε, Σόλτ ε, και τα υπόλοιπα. Αυτό που είναι σημαντικό ε, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από τις συμβαστικές τροπολογίες είναι να λύσουμε τις ε, διαφορές. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά αυτήν την γνωμοδότηση. Να πω όμως δύο λόγια και για την έκθεση Ντάφ γιατί είμαι σκιώδης. Να πω μονάχα ότι θέλω να συγχαρώ τον Άντριου Ντάφ για την προσπάθεια που έχει καταβάλει έτσι ώστε ε, να υποβάλει αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες ενσωματώνουν την θέση του ΕΛΚ, κάποιων μελών του ΕΛΚ ενδεχομένως θα χρειαστεί να κάνουμε έτσι κάποιες μικρές τροποποιήσεις σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες γιατί ορισμένες από αυτές μας δυσκολεύουν αλλά ευελπιστώ ότι θα βρούμε την κοινή διατύπωση. Θα συναντηθούμε άλλωστε μετά από την συνεδρίασή μας εδώ έτσι ώστε να λύσουμε τα θέματα αυτά. Ε, πάντως πρέπει να πω ότι σε γενικές γραμμές ε, πιστεύουμε ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες είναι αρκετά ευρύ, είναι οι συμβιβαστικές τροπολογίες είναι αρκετά έτσι ώστε να ενσωματώσουν και τη δικιά μας θέση και θα αμβληθούν και αυτές οι δύο-τρεις δυσκολίες που έχουμε. Θα τις συζητήσουμε μετά έτσι ώστε ίσως αύριο να έχουμε και την τελική απάντηση όσον αφορά και θέση όσον αφορά αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ για τα σχόλια αυτά. Όσο για το συγκεκριμένο θέμα της εκλογής του Προέδρου του Συμβουλίου αυτού, του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνω να δεχτούμε το συμβιβασμό της Επιτροπής Οικονομικών που μιλάει για, που κάνει λόγο για το ότι το πρόσωπο αυτό θα διοριστεί, θα οριστεί από το Συμβούλιο μετά από λέει μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής και με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μένα το σημαντικό είναι να ακούσουμε, να κάνουμε μια ακρόαση του προσώπου αυτού ή και ατόμου. Γιατί δεν είναι η ίδια διαδικασία όπως για τον ορισμό του ειδικού εκπροσώπου, της υπάτης εκπροσώπου Εκατερίνης Άστον, όπου διορίζεται κάποιος, εγκρίνεται και μετά και μετά παίρνει την άδεια από το κοινοβούλιο να πάει στο αεροδρόμιο να φύγει. Αυτός ο διορισμός πρέπει να γίνει με κάποια πιο συνεπή διαδικασία σαν την παρόμοια με τις έγκρισεις των επιτρόπων. Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε έναν τρόπο διατύπωσης που να το εκφράζει αυτό σαφώς. Αλλά απλή έγκριση από το Κοινοβούλιο όπως προτείνει η Επιτροπή Εικόν είναι κάτι το ασαφές. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το επεξεργαστούμε περαιτέρω. η Οικονομική Επιτροπή θα αναβάλει την ψηφοφορία της μέχρι το Δεκέμβριο, έτσι νομίζω και πιστεύω. Μάλιστα κύριε συνάδελφε, ο κύριος Σεσκόφσκι θέλησε να εκφραστεί επίσης, έχει το λόγο. Κοιτάξτε, δεν έχω τίποτε επαναστατικό να σας πω, απλώς ότι πολλές φορές το θέμα είναι ότι υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά ίσως υπερβάλλουμε το τι μπορούμε να κάνουμε με τις ισχύουσες συνθήκες χωρίς αλλαγές τους. Πρέπει βέβαια να είμαστε φιλόδοξοι και συμφωνώ με τους κύριους συζητητές για το θέμα δε... Όχι για το θέμα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα ήθελαν να συμπεριληφθούν και οι χώρες εκτός Ευρωζώνης αλλά που θέλουν να μπουν σε αυτήν στη, στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο δυνατόν περισσότερες και περισσότερο. Δεν ξέρω άμα γίνεται όμως. Και από τις υπάρχουσες προτάσεις της οίκων του ΝΤΑΦ και άλλων μπορεί να βρεθεί κάποια συνένεση και συμβιβασμός. και να αποφασίσουμε το σωστότερο. Απλώς επιβεβαιώνω ότι συμφωνεί και το ΕΛΚ εκτός από μερικές λεπτομέρειες. Να, αυτά είχα να σας πω. Να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα όσο δυνατόν περισσότερο και να βρούμε μια λύση όπου το Συμβούλιο Επιτήρησης Εποπτείας θα είναι αποτελεσματικό για να είμαστε βέβαιοι ότι θα λειτουργήσουν τα πράγματα όπως θέλουμε. Ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε Κύριε συνάδελφοι όλοι. Αύριο το πρωί στις 10 θα ψηφίσουμε τις δύο αυτές εκθέσεις. Η Επιτροπή Οικονομικών θα αποφάσιζε τέλη Νοεμβρίου, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αυτό. Μπορεί, λέει, να γίνει αναβολή. Λοιπόν, έληξε αυτή η συζήτηση και τώρα περνάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής μας ημερήσιας διάταξης, που είναι συζήτηση για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία περί δημογραφίας. Σας υπενθυμίζω ότι με βάση μια κάπως καθυστερημένη ανακοίνωση της, Κομισιόν, ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος πρέπει να αποφανθούμε σύμφωνα με την διαδικασία κατεπήγοντος. Ό, έτσι συμφώνησαν οι συντονιστές και οι συντονίστριες. Και γι' αυτό έχουμε ήδη εννιά τροπολογίες που κατατέθηκαν από πολλούς συναδέλφους και καλό όσους τις έχουν συντάξει και όσες να μας τις παρουσιάσουν αν θέλουν Υπάρχει κανείς τέτοιος ή τέτοια. Καμιά αποσαφήνιση μήπως θέλετε απορία να λύσουμε. Ο Ανδρέας Νταφ. Είδα τις τροπολογίες του ΕΛΚ και νομίζω ότι μερικές από αυτές δείχνουν ότι υπάρχει παρεξήγηση της φύσης της εκθέσεως αυτής. Η Κομισιόν προσπαθεί να αποσαφηνίσει τα τεχνικά θέματα σε σχέση που αφορούν τη συλλογή δημογραφικών στατιστικών στοιχείων. Και όχι να αλλάξει την ισχύουσα διαδικασία. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τον ορισμό του τι είναι ενισχυμένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο. είναι λάθος αντίληψη αυτό. Παρεξήγηση. Λάθος δηλαδή. Και νομίζω ότι πρέπει να επανορθώσει τα πράγματα ο εισηγητής ή οι συντάκτες των μερικών τροπολογιών μάλλον. Ευχαριστώ άλλος. Αντρέα μήπως δεν κατάλαβα τι εννοούσε όταν μίλησες για λάθος. Να μου το εξηγήσεις πριν σχολιάσω εγώ. Α, όχι εγώ, εγώ. Κοιτάξαμε την ε, διατύπωση πολύ προσεκτικά και μου φαίνεται ότι είπατε ότι κάναμε παρεξήγηση. Δεν νομίζω. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι όσο αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές Μεγάλος αριθμός πολιτών από τις λεγόμενες νέες χώρες μέλη που έχουν εγκατασταθεί στις παλαιότερες θα συμπεριλαμβάνονται τώρα, θα μετρούνται ως ψηφοφόροι του πληθυσμού των παλαιών χωρών μελών. Ξέρουμε ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο Ρουμάνοι ζουν εκτός Ρουμανίας και θα μετρηθούν αλλού. Υπάρχει μεγάλος αριθμός Πολωνών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρόμοιο πρόβλημα. Είναι λοιπόν σημαντικό να το κανονίσουμε αυτό λέγοντας ότι η θαγένεια του κράτους μετράει και όχι η απλή εγκατάσταση. Οι δημογράφοι συμφώνησαν ότι ναι μεν σωστό, θεμητό είναι να εγκαθίσταται κανείς όπου θέλει, αλλά οι υπολογισμοί των ψηφοφόρων πρέπει να γίνουν αλλιώς. Αυτό, σε αυτό βασίζονται οι τροπολογίες μας και δεν είναι παρεξήγηση. Ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, εγώ τώρα διάβασα το σχόλιο της Κομισιόν για την τροπολογία της Επιτροπής ΑΠΑΣΧ και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το διαβάσουμε όλοι. Πρέπει να σας πω ότι ο Ιταλός ή και ο Ιταλός θα είχα συμφέρον να ακολουθήσουμε την αρχή της Ιθαγενείας γιατί τότε θα ήμασταν η πιο πολυπληθής χώρα της Ευρώπης. Αλλιώς. Η λογική όμως της Κομισιόν φαίνεται σωστότερη, δηλαδή να ακολουθείται η συνήθις μέθοδος υπολογισμού. Και αυτό συμφωνεί και με τις συστάσεις του ΟΗΕ για τη 12μηνη περίοδο. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Ο κανονισμός καθορίζει απλώς ένα κοινό πλαίσιο για τον τρόπο εφαρμογής ορισμένων κανόνων. Πρέπει επίσης να σας πω ότι και για τον, την κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο δεν χρησιμοποιείται η ηθαγένεια αλλά η κατοικία. Μπορούμε αν θέλουμε βέβαια να αλλάξουμε το κριτήριο. Όπως σας είπα, αν είναι με το κριτήριο της κατοικίας θα έχουμε πολλά ωφέλη εμείς η Ιταλία, αλλά ε, με το κριτήριο της Ιταγένης μάλλον. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει τέτοια μεγάλη αλλαγή. Η πρόταση της Κομισιόν γενικότερα μου φαίνεται πιο λογική και πιο σύμφωνη με την ισχύουσα διαδικασία. Καζόφσκι. Εγώ το έχω μελετήσει το πρόβλημα. Αυτά που λέτε εσείς και η Κομισιόν είναι σαν να υπάρχει status quo που δεν αλλάζει και ότι είναι καινούργια η ιδέα να αλλάξει το κριτήριο σε κριτήριο ηθαγένειας αλλά τώρα υπάρχει δυνατότητα να ορίζουν οι χώρες μέλη τι εννοούν με την έννοια εγκατάσταση. Μερικές φορές ορισμένοι κάτοικοι χωρών είναι εγγεγραμμένοι, άλλοι όχι. Και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτό. Εμείς βασιζόμαστε στην ευελιξία, δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη θα δηλώσουν οικειοθελώς τον αριθμό των κατοίκων ενώ τώρα δημιουργείται μια νέα κατηγορία, δηλαδή συνήθις κατοικία, δωδεκάμινη, διάρκεια κλπ. Και αυτό είναι δύσκολο να καθοριστεί το κριτήριο, να εφαρμοστεί μάλλον. Άρα καταλήγουν ότι για το Eurostat και την Κομισιόν το κριτήριο της συνήθους κατοικίας θα εφαρμοστεί αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και το σύνηθες κριτήριο που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα. και θέλουν να επιμείνουν σε αυτή τη νέα κατηγορία της συνήθους κατοικίας που είναι δύσκολο να καθοριστεί και θα δημιουργούσε και όλα τα προβλήματα που ανέφερε και ο Γκιόργη πράγμα λεπτό για ορισμένες χώρες μέλη γιατί δεν έχει γίνει καμία μελέτη και η Κομισιόν μας λέει θα κάνουμε προσωμιώσεις για να δούμε αν μπορεί αυτό το κριτήριο της συνήθους κατοικίας να εφαρμοστεί. Α, δεν έχουν γίνει. Ούτε τι επιπτώσεις θα είχαν αυτά τα κριτήρια. Γι' αυτό υποστηρίζω την ιδέα ότι δεν πρόκειται για παρεξήγηση. Δεν λέω να υποστηρίξουμε τις πιο ακραίες αποφάσεις και να αλλάξει το κριτήριο τελείως και να περιορίζεται μόνο στην ηθαγένεια. Αλλά μέχρι τώρα υπήρχε η ευελιξία και δεν χρειάζεται νέα κατηγορία που δεν έχει δοκιμαστεί και που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον τρόπο των υπολογισμών. Προσθέτω δε ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στην τελευταία έκθεση του Βαν Ρόμποϊ για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των δημοσιονομικών. Και πάλι είναι ασαφές πώς θα χρησιμοποιηθούν εκεί τα στατιστικά δεδομένα, κατηγορία 1 με ευελιξία ή κατηγορία 2 χωρίς ευελιξία, όπως ζητάει το Συμβούλιο. Να το προσέξουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφός μας Χέφνερ. Yes, thank you. Well, to... Ναι, ευχαριστώ. Στα αγγλικά. Θα είμαι σύντομος. Ούτε εγώ βλέπω τα πλέον εκτίματα της αλλαγής αυτής. Αντίθετα βλέπω να αναδύονται νέα προβλήματα. Στις συνθήκες έχουμε νέες κατηγορίες τώρα και ε, νέους πληθυσμούς που θα οδηγήσουν και σε τεχνικά ζητήματα έτσι ως προς τη δημογραφία. Χρειάζεται μεγάλη ανταλλαγή δεδομένων και τα λοιπά. Και ανοίγουμε τώρα τους ασκούς του αιώλου. Και δεν καταλαβαίνω και το σκεπτικό που κρύβεται από πίσω. Και πραγματικά ας παραμείνουμε στον πληθυσμό αυστηρά και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Βίλαντ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι αυτή την όλη συζήτηση ότι θεωρώ έτσι κάπως εκπληκτική. Αυτή η όλη ιστορία είναι της Επιτροπής Απασχόλησης. Καλό θα, εντάξει, θα καταλαβαίνω αυτό αν ήταν στατιστικές για την αγορά εργασίας. Αλλά μπαίνουν στα δικά μας καθημερινά χωράφια. Δεν κατάλαβα γιατί σε αυτό το θέμα ε, ε, επί της ουσίας αρμόδια δεν είναι η δική μας επιτροπή και είναι η Επιτροπή Απασχόλησης. Είπαμε κάθε αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο πιο αδύναμος κρίκος της. Έχουμε ε, στο Κοινοβούλιο νομοθεσία, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και ε, νομιμοποίηση και μπορεί να κάνουμε όσο θέλουμε με ακρίβεια τα πράγματα εάν χωλένουμε σε τέτοιες περιπτώσεις τότε και η υπόλοιπη αλυσίδα είναι το ίδιο νεπαρκής όσο είναι αυτός ο κρίκος της. Λοιπόν, Και πραγματικά αυτοί οι κύριοι που φτιάξαν τις συνθήκες με τα δημογραφικά τα έχουν λίγο μου σκέψει για να το πω έτσι, θαλασσώσει. Και ό,τι έχει να κάνει ε, με την προσώπηση και αντιπροσώπευση ε, θα πρέπει να συνδέεται με εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου όπως ισχύει σε κάθε κράτος μέλος για την εσωτερική ενόμη τάξη. Δεν είναι όσοι ζουν σε μια χώρα, ε, δεν έχουν όλοι το δικαίωμα του εκλέγην. Και σε κάθε εκλογή μία ψήφο έχει ο καθένας. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια κατανομή. Προς το παρόν αισθάνομαι περίεργα και δηλώνω αδυναμία να το μελετήσω αυτό το θέμα σε βάθος. Και αυτό είναι ένα εργοτάξιο που γίνονται χοντρά έργα. Και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι για πει. Πρέπει να το ρυθμίσουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τα αφήσω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ρυθμιστεί. Ε, ε, ό,τι υπερβαίνει την αμυγή στατιστική της αγοράς εργασίας θα πρέπει το συντομότερο να έρθει εδώ και όχι στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφοι, ο κύριο Μπρόν, ζήτησε το λόγο. Yes, I'm, I'm less... Δεν με απασχολεί τόσο πολύ η, η στατιστική μέθοδος, με απασχολεί περισσότερο η ουσία και το θέμα των στατιστικών. Στην έκθεση αναφέρεται ε, αναφέρονται μάλλον ε, οι ε, αυξανόμενες προκλήσεις δημοκρατικές, αναφέρονται τα ποσοστά γονιμότητας και δίνονται και κάποια στοιχεία σχετικών πληθυσμών. Δεν γίνεται όμως καμία αναφορά στις μαζικές αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα εδώ τα τελευταία 60 περίπου χρόνια ε, στην προέλευση των ε, πληθυσμών, κυρίως στις μεγάλες ε, πόλεις της Δυτικής Ευρώπης. Στην Ανατολική Ευρώπη ακόμα δεν έχει αρχίσει αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι στο αναφέρεται και στο, στη διαδικασία 2020 ότι ε, θα ε, πρέπει να ε, μπουν νέα εργατικά χέρια γιατί υπάρχει φθήνουσα δημογραφία στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να δεχτούμε τέτοια πράγματα. Γυράσκει ο πληθυσμός της Ευρώπης ε, και ε, ε, τελικά αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι είναι να φεύγουν και να αλλάζουν τόπο διαμονής και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τελικά καμία συζήτηση για το κατά πόσον οι πολίτες μας θέλουν τις αλλαγές αυτές. Βλέπω ότι στο έγγραφο εδώ γίνεται λόγος σε σημαντική διάσταση μίσους που μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι δημογραφικές στατιστικές. Ευχαριστώ αγαπητές, αγαπητές συνάδελφοι. Δεν νομίζω ότι ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ κυρία Κλεμανσό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να πει ότι ε, χαίρεται γιατί βλέπει ότι οι περισσότεροι μεταξύ ημών στηρίζεται την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δημογραφικές στατιστικές γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, συμφωνήσουμε επί της κοινή βάσης των ευρωπαϊκών στατιστικών στη δημογραφία. Με τον κανονισμό αυτό έχουμε δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να ορίσουμε και να δημιουργήσουμε μία βάση για σταθερές, για ε, ε, περιοδικές στατιστικές, ε, οι οποίες όμως θα φτάνουν σε ικανό βαθμό λεπτομέρειας. Flexibility. That means ε, θα θέλαμε όμως εδώ ε, να προσθεθεί και η ιδέα ε, του, της συνήθους διαμονής και του συνήθως διαμένοντος. Αυτό είναι σημαντικό γιατί επίσης ο άλλος μεγάλος στόχος της ψηφοφορίας με ε, κατά πλειοψηφία, με ενισχυμένη πλειοψηφία, δεν μας δίνει το δικαίωμα ε, να επιτρέψουμε την πλήρη ευελιξία, γιατί η πλήρης ευελιξία θα δημιουργήσει προβλήματα ε, γιατί ας πούμε θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά τους ε, Ρουμάνους ε, που καταγράφονται όχι μόνο στην Ρουμανία αλλά και στην Ιταλία και στην Ισπανία κλπ. Επομένως δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε την κατάσταση ως έχει. Γιατί έτσι αφήνουμε περιθώριο για διπλό, για διπλό υπολογισμό, για διπλή μέτρηση των πληθυσμών αυτών. Θέλουμε λοιπόν Λοιπόν να είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά τον ορισμό. Τώρα, ποιο είναι ο ορισμό ο οποίο ε, θα χρησιμοποιηθεί. Έχουμε ε, μια εσωτερική ε, σύσταση, σύσταση, η οποία όχι μόνο στην Ευρώπη και σε διεθνέ παγκόσμιο επίπεδο έχει συζητηθεί επί μακρόν. Μετά από πολιετής συζητήσεις λοιπόν έχουμε πλέον ορισμό ε, που βασίζεται ε, στην, στο κριτήριο αυτό των 12 μηνών ε, τόπος συνήθους διαμονής με αυτήν την 12 μηνή διάρκεια. Τώρα το θέμα της ηθαγένειας, δηλαδή ο ορισμός ο οποίος βασίζεται στην ηθαγένεια, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ σε διεθνές επίπεδο τεχνικά ε, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο γιατί αυτό θα προϋπέθεται ανταλλαγή δεδομένων σε εθνικό επίπεδο ε, και δεν νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Πραγματικά δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν από τεχνικής απόψεως αμφιβάλλουμε πολύ ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε να παραμείνουμε σε, αυτόν τον ορισμό της συνήθους διαμονής 12 μήνης διάρκειας. Και μπορούμε επίσης να πούμε ότι αυτό ευθυγραμμίζεται με άλλους κανονισμούς που έχουν ε, εγκριθεί προηγούμενα ε, όσον αφορά τις στατιστικές μετανάστευσης κλπ. Επομένως και για λόγους συνεκτικότητας θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτόν τον ορισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα, σύντομα. Εγώ το πρόβλημα που βλέπω είναι το εξής η εκπροσώπηση είναι πολιτική κατηγορία και νομίζω ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί ή να οριστεί αλλιώς από δημογραφικό βόλο για να βολευτούμε δημογραφικά. Γιατί αλλιώς θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου υποθετικά θα έχουμε Βρετανούς ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπούν Πολωνούς, Ισπανούς ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπούν Ρουμάνους κλπ. Μπορεί να γίνεται, αλλά έχω αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον γίνεται. Και τότε θα ξαναγυρίσουμε στην ιδέα του Ευρωπαϊκού Μητρώου. Θυμάστε ότι μερικοί το είχαν προτείνει για τα πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια. Είναι δύσκολο. Αλλά αν μιλάμε για ευρωπαϊκή ηθαγένεια, τότε πρέπει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό Μητρώο. Ζητώ συγγνώμη πρώτα απ' όλα για την ε, μακρά μου ε, απουσία. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Ο Τλάνφος Ταρκόφσκι και μετά ο κύριος ε, Νταφ. Δεν θυμάμαι να έχω διαφωνήσει με τον Γιώργη, αλλά εδώ έχω πρόβλημα δεν με προβληματίζει τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί τουλάχιστον όταν ε, μιλάμε ας πούμε, ε, για την αντιμετώπιση της, συνθήκης του, αντιμετώπιση της, εθνικής, ε, της ευρωπαϊκής από τη συνθήκη του Μάστερ και δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου ας πούμε, εκπρόσωποι, όπου μπορούσαν οι Ισπανοί οι βουλευτές να εκπροσωπούν ε, τους συνήθως διαμένοντες στην ε, Ρουμάνους ας πούμε. Αλλά έχω ένα πρόβλημα όμως όσον αφορά ε, ε, το Συμβούλιο, την εκπροσώπηση ε, στο Συμβούλιο. Εκεί βεβαίως η λογική βασίζεται στην ηθαγένεια. Και δεν έχουμε, δεν παρουσιάζει το σύστημα αυτή την ευελιξία. Αυτό με απασχολεί και επίσης όταν συζητάμε ένα ζήτημα το οποίο ανέφερα και προηγουμένως, δηλαδή εάν θα έχουμε ας πούμε ενδιάμεση αναθεώρηση στον προϋπολογισμό και εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε την δυνατότητα ε, να ε, δώσουμε, ε, να έχουμε ένα άνοιγμα προς τα εθνικά επιδόματα, εκεί θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα. Έχει κάνει καμιά μελέτη προσωμείωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ε, ξέρει επίσης πώς θα κατευθυνθεί η ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάφα. Κοιτάξτε, το εξέτασα βέβαια όταν συντάσαμε, όταν συνέτασα τις εκθέσεις μου για τα διεθνικά ψηφοδέλτια. Υπάρχουν βέβαια 27 διαφορετικές και αντιφατικές μεταξύ τους, ε, διαφορετική και αντιφατική μεταξύ τους ορισμοί της ηθαγένειας. Δεν είναι ενιαίο το σύστημα. ώστε να πούμε ότι μπορεί να αρχίσει εύκολα να υπάρχει, να εφαρμόζεται ένας ενιαίος ορισμός της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Πολύ πρακτικότερο και λογικότερο θα ήταν να περιοριστούμε στη συνθήκη, στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δημογραφικά στατιστικά στοιχεία όπου που ακολουθούμε ως συνήθως. Δεύτερον, η συνθήκη περιγράφει, ορίζει την ενισχυμένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο ως βασιζόμενη στον πληθυσμό και όχι στην ηθά γένεια. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει τη γνωμοδότηση να τη θεωρήσουμε ως σημαντική μεν αλλά τεχνική. Συμφωνώ όμως απόλυτα με τον κύριο Βίλαντ ότι παράλογο είναι η Επιτροπή Απασχόλησης να είναι η κύρια Επιτροπή Αρμόδια επί της ουσίας εδώ. Mm. Πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, βλέπω ότι ήδη έχει σηκώσει το χέρι του συνάδελφος ε, Γκουελτιέρη και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, Γκουελτιέρη, πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Πρέπει και εγώ να πω ότι στηρίζω αυτό που είπε ο συνάδελφος Βίλεντ. Την άποψή του δηλαδή ότι είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι η αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Απασχόλησης, μια και ε, το ζήτημα παρουσιάζει ε, τόσο ε, έντονα πολιτικά και θεσμικά ζητήματα τα οποία άπτονται των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 4, τουλάχιστον το άρθρο 4, θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα της ΑΦΚΟ. Εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας. Εκτιμώ την προσπάθεια πολιτικής διαμεσολάβησης του Ράφα. Αλλά από άποψη ρεαλιστική και ορθολογική. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν η ευελιξία οδηγήσει στο γεγονός ότι δύο φορές θα προσμετρώνται οι ίδιοι άνθρωποι, τότε οδηγούμεθα στο, στη διαπίστωση πρέπει να υπάρχει ένα ομοιογενές κριτήριο. Εάν αυτό το ομοιογενές κριτήριο ε, είναι η ηθαγένεια ή τι να σας πω, τότε θα πρέπει να πούμε ας πούμε ότι μια χώρα έχει περισσότερους πολίτες από τους άλλους, από, μια άλλη χώρα. αλλά δεν νομίζω ότι όλοι θα ε, συμφωνήσουν ότι ας πούμε η Ιταλία είναι η πιο πολυπληθής νέα χώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βασιστούμε στα διεθνή ε, στάνταρ, στα διεθνή πρότυπα και ότι ο καθένας ε, προσμετράται μία φορά και όχι δύο. Αυτό είναι το πιο λογικό. Το πρόβλημα της ευελιξίας, αν, το ζήτημα μάλλον της ευελιξίας, αν οδηγήσει σε τέτοιες μεγάλες διαφορές, θα μπορούσε να, θα μπορούσε να ε, δυναμητήσει την αξιοπιστία αυτού του τρόπου υπολογισμού. Και επομένως ρωτώ και εγώ, μήπως μπορούμε να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, έτσι ίσως να επαναδιαπραγματευτούμε το ποιος θα είναι, ποια επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό. Διαφορετικά, λογικά, και πολιτικά η πρόταση της Κομισιόν είναι η πιο δυνατή. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, η κυρία Κλεμασό παρακαλώ να μας δώσει μια νέα απάντηση υπό το φως των νέων ερωτημάτων που έχουν τεθεί. Yeah, thank you very, very Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν νέα στοιχεία. Μόνο το ερώτημα για την ε, προσωμείωση, αν έχουν υπάρξει προσωμιώσεις. Όχι. Η απαντήση είναι όχι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακριβείς προσωμιώσεις, γιατί σε πολλές χώρες ε, πρέπει ακόμα να γίνει κάποια δουλειά, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε ε, σε, αυτήν, σε αυτόν τον ορισμό των ε, συνήθως διαμενόντων με το κριτήριο των 12 μηνών. Γνωρίζουμε πάντως ε, ότι θα γίνει αυτό. Ε, εν εγώ έδωσα το παράδειγμα της Ρουμανίας και είναι σαφές ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει επίπτωση, αλλά και σε άλλες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω λοιπόν ότι ε, αυτό το ζήτημα θα απασχολήσει και την συνεδρίαση των συντονιστών η οποία θα ξεκινήσει ως ονούπο. Θα συζητηθεί λοιπόν, θα σταματήσουμε ε, τα διακλεπτά θα ολοκληρώσουμε την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής και σε πέντε λεπτάκια ξεκινούμε και την συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ.